Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχει web streaming για τη σημερινή συνεδρίαση από 6 μέχρι 6.30 σε σχέση με την προετοιμασία της αντιπροσωπείας στην Ελλάδα. Θα, για τις 27 με 29 Απριλίου θα γίνει μια ακρόαση των ε, υπαλλήλων της Όλαφ και κλεισμένων των θυρών μπορούν να παραμείνουν μόνο οι βουλευτές δηλαδή στην αίθουσα και μέλη της γραμματείας. Όλοι οι άλλοι θα πρέπει να αποχωρήσουν. Στις 6 τα πρακτικά της 15ης-16 Μαρτίου 2010 έχουν αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 7 Απριλίου. Περνάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης που είναι η ειδική έκθεση 18 κάθετος 2009 του ελεγκτικού συνεδρίου σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της στήριξης του ΕΤΑ για την περιφερειακή και οικονομική ολοκλήρωση στην Ανατολική Αφρική και τη Δυτική Αφρική. Δίνουμε το λόγο στον κύριο Κίνς, τον εκπρόσωπο του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω κάπως σύντομα την έκθεση 18-2009 του Ελεκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την στήριξη της περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης στην Ανατολική Αφρική και την Δυτική Αφρική. Στο έγγραφό του, ο κύριος Στάς, ο εισηγητής, συνοψίζει πολύ καλά τις παρατηρήσεις του λεγκτικού συνεδρίου, τα συμπεράσματά του και τις συστάσεις του. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι αυτό που θα έπρεπε να κάνω εγώ τώρα είναι να υπογραμμίσω τα εξή. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την στήριξη για την περιφερειακή οικονομική ολοκλήρωση στις δύο αυτές περιοχές, έχει επιτευχθεί εν μέρη για διάφορους λόγους. Ορισμένοι από αυτούς δεν εξαρτώνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως για παράδειγμα ότι υπάρχει μια πληθώρα περιφερειακών οργανώσεων που πολλές φορές επικαλύπτονται. Δεύτερον, όσον αφορά τις απαντήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι συστάσεις, η σύσταση αριθμός 1 στην παράγραφο 57 της έκθεσής μας που αναφέρεται στο διάλογο με τις περιφερειακές οργανώσεις λέει ότι είναι προς όφελος της περιφερειακής ε, ολοκλήρωσης εν ώψη της Συμφωνίας Κοτονού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως θα πρέπει να αποφασίσει και να φροντίσει να πάρει μέτρα για πιο αποτελεσματική και καλύτερη απόδοση των κονδυλίων ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξη. Επίση, η Συμφωνία Κοτονού λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίση την ευθύνη για οικονομικέ αποφάσει υπέρ της ε, χρήσης κονδυλίων του ΕΤΑ. Τρίτον, όσον αφορά τη δικιά μας σύσταση αριθμό 2, που αναφέρεται σε περισσότερη συνοχή ανάμεσα στη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την περιφερειακή αλλά και εθνική στρατηγική. Πρέπει να υπάρξει στρατηγική σε εθνικό επίπεδο και η περιφερειακή ολοκλήρωση και σχετικές συμφωνίες συχνά υστερούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή της είχε υποσχεθεί να ασχοληθεί με το θέμα αυτό κατά τη μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση του ΕΤΑ, αλλά υπάρχει ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναφέρει τα προκαταρκτικά αποτελέσματα αυτής της ενδιάμεσης ε, αξιολόγησης που δεν συμπεριλαμβάνει όμως το στοιχείο αυτό. Τέλος, θέλω να αναφερθώ στα ποσά που δίνονται για την περιφερειακή συνεργασία, που είναι δύο φορές το ποσό που δίνεται βάσει του ένατου ετά. Τώρα στο δέκατο έχουμε περίπου το διπλό ποσό, διότι είχαμε στο ένατο 904 εκατομμύρια και με το δέκατο ετά 1783 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν οικονομικές ε, συμφωνίες οι οποίες όμως δεν προχώρησαν όπως είχα προβλεφθεί. Έτσι υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Υπάρχει αδυναμία στην ε, απορροφητική ικανότητα των περιφερειακών οργανώσεων που τις κάνει να μην μπορούν αποτελεσματικά και αποδοτικά να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια αυτά. Τέλος κύριε Πρόεδρε, θέλω να εκφράσω εδώ την εκτίμηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχτηκε τις περισσότερες από τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Κίνστε. Έμαθα ότι ο κύριος Μπάρτ Στάις δεν είναι παρόν γιατί είναι άρρωστος, άρα νομίζω ότι θα πρέπει σε μια προσεχή συνεδρίαση να δώσουμε τη δυνατότητα στον κύριο Στάς να παρέμβει ως εισηγητής και να προσθέσει κάτι σε σχέση με αυτά που προανέφερε το Ελληνικό Συνεδρίο, κύριε Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του, στον κύριο Στάς. Ενδιαφερόμαστε να δούμε τα συμπεράσματά του, τα οποία δεν υπάρχουν ακόμη. Μάλλον ε, περαστικά ευχόμαστε τον κύριο ε, Στάς. Ε, ε, ζητούμε Δεν έχουμε τα συμπεράσματά του λοιπόν ακόμα. Τώρα, η, η Κομισιόν χειρίζεται το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο και για λογαριασμό των χωρών μελών και εμείς έχουμε περιορισμένη επιρροή σε αυτό. Τα χρήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά, να έχουμε δηλαδή διαφορετικά αποτελέσματα από άλλους τομείς της αναπτυξιακής βοήθειας με χρήματα που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από άλλες πηγές. Εξετάζοντας τα όσα έχετε σημειώσει εδώ, δεν βλέπω διαφορά. Μπορώ να θέσω τότε και το θέμα της εγγραφής στον προπολογισμό του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αναπτύξεως. Διότι οι χώρες μέλη εφόσον κάτι τι είναι σημαντικό και έχει πολιτική προτεραιότητα, το κρίνουν διαφορετικά και αυτό θα πρέπει να εμφανίζεται και εδώ. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε τώρα, κύριε Κίνστα. Ίσως καλύτερα να μου υποβάλλετε πρώτα όλες τις ερωτήσεις και θα απαντήσω μια και καλή. Η κυρία Γιάλα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κίνης μερικά πράγματα, αφού προηγουμένως τον ευχαριστήσω για την έκθεσή του και να ευχηθώ και εγώ περαστικά στον κύριο Στάς. Επειδή συμμετέχω και στην Επιτροπή Μεταφορών, με ενδιαφέρει πολύ αυτά που λέει η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου σχετικά με τον μόνο τομέα από ό,τι λέει όπου μπορέσαν να επαληθεύσουν την ε, προσπάθεια περιφερειακής ε, ολοκλήρωσης στην περιοχή ήταν ακριβώ ο τομέας των μεταφορών. Θα ήθελα λοιπόν ο κύριος Κίνης να μπει κάπως περισσότερο σε βάθος. Δηλαδή ποια είναι τα θετικά από την βοήθεια αυτή στις μεταφορές, μήπω την εμπειρία αυτή μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε και σε άλλου τομείς. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, δίνω το λόγο στο ελεγκτικό συνέδριο, στον εκπρόσωπό της. Παρακαλώ κύριε Κίνστα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Για την πρώτη ερώτηση της κυρίας Γκρέσλε δεν είχε άμεση σχέση με τον προπολογισμό του ΕΤΑ ή με τον καλύτερο έλεγχο και τις δαπάνες. Το ελεκτικό συνέδριο έχει πει ότι στηρίζει την έκφραση αυτή του προπολογισμού, αλλά τα προβλήματα τα, μία, οποία εμεί αναφέρουμε στην έκθεσή μας δεν έχουν να κάνουν τόσο με τον έλεγχο των ποσών. Έχουν να κάνουν με διάφορα ζητήματα οργάνωσης κυρίως. Μερικά έχουν να κάνουν με τον προπολογισμό, με τα νούμερα. Οι περιφερειακές πτυχές της συνεργασίας αυτής, για παράδειγμα, δεν εμφανίζονται στο εθνικό επίπεδο. Σημειώσαμε επίσης και κάποια άλλα προβλήματα. Την ικανότητα απορρόφησης των περιφερειακών οργανώσεων, της καθυστερήσεις των προγραμμάτων και αν δείτε πόσα προγράμματα ήταν αποτελεσματικά και πόσα είχαν αδυναμίες, θα δείτε. Γιατί λέμε ότι οι στόχοι μας δεν έχουν επιτευχθεί μόνο 6 ή 5 από τα 18 προγράμματα, έστω και μερικώς έφεραν κάποια αποτελέσματα. Τα υπόλοιπα αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες. Τέλος, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στην περιφερειακή ολοκλήρωση δεν έχουν να κάνουν τόσο πολύ με το γεγονός ότι έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΑ τα προγράμματα αυτά και όχι από τον προϋπολογισμό αυτό καθεαυτό. αυτό. Uh, όσον αφορά τώρα την ερώτηση της κυρίας Αγιάλα, Στην παράγραφο 20 της έκθεσής μας αναφερόμαστε σε αυτό. Ότι οι μεταφορές όσον αφορά την περιφερειακή ολοκλήρωση έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Οπότε έτσι νομίζω ότι απαντάω. Ευχαριστώ. Ζήτησε το λόγο ο κύριος Κουίνς, ε, διευθυντής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω Καταρχήν, ότι η περιφερειακή οροκλήρωση ε, είναι ένα από τα πιο περίπλοκα προγράμματα που διαχειριζόμαστε και η εφαρμογή είναι προβληματική και πιο βραδία από τα εθνικά προγράμματα, διότι έχουμε να κάνουμε ένα ευρύ φάσμα χωρών που έχουν αποκλίνοντα συμφέροντα και περιφερειακές, πολλές περιφερειακές οργανώσεις και όπως ε, πολύ σωστά αναφέρει το ελεγκτικό συνέδριο, υπάρχουν ε, επικαλύψεις ως προς την γεωγραφική συμμετοχή περιφερειακών οργανώσεων και της εντολής τους. Επίσης είναι γεγονός ότι οι περισσότερες περιφερειακές οργανώσεις είναι σχετικά αδύναμες ως προς την διαχείριση και τη δυνατότητα απορρόφησης. Άρα εργαζόμαστε σε έναν πολύ δύσκολο τομέα. Η Επιτροπή καλωσορίζει αυτή την έκθεση, όπως είπε ο κ. Κλίνστ, δεχτήκαμε τις περισσότερες συστάσεις και εκεί που δεν τις δεχτήκαμε είναι θέμα ίσονος σημασίας και όχι ουσίας. Να δούμε τα τρία σημεία που έδειξε ο κύριος Κίστ, Κλίστ. Θεωρούμε ότι χρειαζόμαστε πιο αποδοτικό διάλογο. Οι αποστολές στα τέλη του 2008-2009 ε, ήταν αποτελεσματικές και έκτοτε είχαμε συναντήσει με κάθε περιφέρεια το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ε, ε, πέρυσι, όπου είχαμε μία δήλωση στην περίπτωση της Ανατολικής και μία της Δυτικής Αφρικής, όπου βλέπουμε την ανάγκη των περιφερειών να ασχοληθούν με θέματα τα οποία ε, θίγησαν και από την ε, έκθεση του Λεγκτικού Συνεδρίου, δηλαδή να ε, συντάξουμε έναν οδικό χάρτη για περιφερειακή ολοκλήρωση και μέσα στα πλαίσια του 10ου ΕΤΑ. Επειδή η κυρία Αγιάλα αναφέρθηκε στο θέμα των μεταφορών, θα ήθελα να σας πω ότι πέρσι ε, όλοι οι Υπουργοί Μεταφορών ε, της Δυτικής Αφρικής φτάσαν σε μία δήλωση Μπουρκίνα Φάσο. Είχαμε πολλές δηλώσεις από ό,τι φαίνεται και έτσι ασχοληθήκαμε με το θέμα των υπερφορτωμένων φορτηγών που φαίνεται ε, μικρό θέμα αλλά είναι σημαντικό στη Δυτική Αφρική. Και τώρα έχουν αναλάβει δράσεις επί του θέματος, γιατί αυτό είναι ένα μείζον περιφερειακό πρόβλημα που πλήττει όλο το δίκτυο μεταφόρων. Θα πρέπει λοιπόν να προβάλλουμε τον περιφερειακό διάλογο όπου μπορούμε. Δεύτερον, το θέμα των ενδιάμεσων ε, αναθεωρήσεων. Η Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη συνοχή μεταξύ του τι κάνουμε σε εθνικό επίπεδο και σε περιφερειακό. Η Επιτροπή ανέλαβε αυτό το ζήτημα και θα το δούμε και στην ενδιάμεση, εθνική ενδιάμεση αναθεώρηση των κρατών και θα αρχίσει του χρόνου το ενδιάμεσο πρόγραμμα αναθεώρησης. Άρα θα ληφθεί υπόψη και δέχομαι αυτά που είπε και ο κύριος ε, Κλίν στο έγγραφο, διότι δεν υπάρχει τελική έκβαση ως προς τη... τον προγραμματισμό. Ως προς την αύξηση των περιφερειακών προγραμμάτων, όπως είπε ο κύριος Κλίνστ, έχουμε ε, έναν διπλασιασμό του 10 του προγράμματος σε σχέση με το 1ο. Είναι μεγάλη η πρόκληση, αλλά σχετίζεται και με την ανάγκη επιτάχυση της διαδικασίας και βεβαίως και να ε, ενισχύσουμε τα ΕΠΑ. Άρα έχει προωθηθεί ο διάλογος μεταξύ των βασικών ε, περιφερειακών οργανώσεων, την, ε, την ΣΑΝΤΕΚ, την ΚΟΜΕΣΑ και την την οργάνωση της Ανατολικής Αφρικής για να προβάλλει τις δικές της προτάσεις, να εμβαθύνουμε δηλαδή την ε, περιφερειακή ολοκλήρωση στη Δυτική και Ανατολική Αφρική. Άρα έχουμε προβάλει και την ε, οικονομική πρόταση, την οικονομική πρόταση εταιρικότητας έτσι ώστε να ενταχθεί στον οδικό χάρτη. Τα περιφερειακά προγράμματα είναι περίπλοκα και δυνάμει του δεκάτου έτα έχουμε ένα 1% της χρηματοδότησης στην Ανατολική Αφρική όπου τα πράγματα έχουν αλλάξει άρδιν. Μετά τις αποστολές του ελεγκτικού έχουμε υποχρεώσεις 20% και έχουμε ένα βασικό πρόγραμμα το οποίο εξελίσσεται πέρσι εξελίχθηκε πέρσι και φέτος. Άρα προωθούνται οι συζητήσεις και με τις ε, δύο περιφέρειες, γνωρίζουν τι ανέφερε το ελεγκτικό και θα συνεχίσουμε το διάλογο με τις ε, χώρες και τις περιφέρειες όσο προχωράμε. Ευχαριστούμε, Γκέιερ. Ευχαριστώ. Ερώτηση προς τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εξετάζοντας τις έκτακτες εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου σχετικά με εξωτερικές βοήθειες, άλλωστε εμείς κάναμε τη σχετική κριτική στην έκθεση περί απαλλαγής, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλά σφάλματα τα οποία εξηγούνται στην έκθεση ή στην δήλωσή σας αν θέλετε που μας είπατε που μας δώσατε πριν είπατε ότι δεν υπάρχουν στόχοι για την απορροφητικότητα των ε, χωρών αυτών. Πώς μετρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν να προωθηθούν τα προγράμματα αυτά την δυνατότητα διαχείρισης και απορροφητικότητα των χωρών αυτών. Γιατί στη βάση αυτή πρέπει βεβαίως να διαμορφωθούν τα προγράμματα. Η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Με θίγει η κριτική του ελεγκτικού συνεδρίου για την έκθεση αυτή, διότι θίγει και τα θέματα εκείνα όπου και εμείς διαπιστώνουμε προβλήματα στο συντονισμό στους κόρπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό βεβαίως δεν είναι υπέρ ούτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και γι' αυτό επιμένω ότι η κριτική αυτή είναι εξαιρετικά δυσάρεστη έχουμε κατακαιρματισμένη αρμοδιότητα μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα προσθεθεί άλλη μια οργάνωση τώρα. Τότε πραγματικά επιδεινώνονται οι φόβοι μου. Πώς θα βρεθεί η διέξοδος. Είναι πολύ δύσκολο. Το ερώτημα δηλαδή, τι θα κάνουν οι αντιπροσωπείες και τι θα κάνει το κεντρικό όργανο για να κατευθύνει τι αντιπροσωπείες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, γιατί ήδη από το 2000 οι αντιπροσωπείες στελεχώνονται με σημαντικό δυναμικό και έχει αυξηθεί το δυναμικό αυτό ήδη κατά 140%. Σημειώνονται λοιπόν επιφυλάξεις εάν το αεροσκάφος διαθέτει πιλότο που να γνωρίζει και πώς να το κατευθύνει στη σωστή κατεύθυνση. Να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν σε ποια συμπεράσματα καταλήγει για τις αντιπροσωπείες και για την κατεύθυνσή τους από το κεντρικό όργανο και αν υπάρχει κάποιος μηχανισμός συντονισμού μεταξύ των αντιπροσωπιών. Δεν λέω τίποτα βέβαια, αλλά ήδη οι επικεφαλής των αντιπροσωπιών συναντώνται τακτικά για να συζητήσουν και με τους desk officers της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ποια είναι τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν λοιπόν. Και διαβάζοντας τις λίγες εκθέσεις που λαμβάνουμε από τις αντιπροσωπίες, είναι λίγες, διαπιστώνουμε, για παράδειγμα σε μια έκθεση λέει ότι τα πρόσωπα στις αντιπροσωπείες, οι δικοί μας, οι Ευρωπαίοι δηλαδή, κατά 40% του χρόνου εργασίας τους είναι απόντες. Είτε διότι βρίσκονται σε εκπαίδευση, είτε διότι έχουν ιδιαίτερα γενναιόδορες ρυθμίσεις για τις διακοπές και ούτω καθεξής. 40% λοιπόν είναι ελεύθερος χρόνος. Εγώ κατέθεσα γραπτή ερώτηση. Η γραπτή αυτή ερώτηση η οποία απαντήθηκε με τα γνωστά μπλα μπλα. Είναι πράγματα λοιπόν όπου οφείλει κανείς να θέσει ερωτήσεις. Ποια είναι τα συγκεκριμένα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν και αν δεν καταλήγουν σε κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα τότε θα κληθούμε εμείς να συναγάγουμε κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα. Διότι θίγεται πλέον ο ίδιος ο πυρήνας του management. Και εμείς καλούμεθα μετά να τα εκπροσωπήσουμε αυτά προς τα έξω. Η κυρία Σέντερ, Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω λίγο να επιμείνω να απευθυνθώ στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα τον ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσε για το πώς δηλαδή οι συμφωνίες οι πιο περιφερειακές όσον αφορά τις μεταφορές, πώς έχουν ε, τεθεί σε εφαρμογή. Αλλά θα ήθελα να πάμε και λίγο πιο μακριά. Έχουμε τη δήλωση της Μπουργκίνα Φάσο. Προχωράμε σε μία εντός εισαγωγικών εναρμόνιση. Θα ήθελα να ξέρω ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ποιος είναι ακριβώς. Τι νέο σύστημα εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να στηρίξει την περιφερειακή συνεργασία σε αυτό το τομέα. Δεύτερον, η Επιτροπή μας λέει ότι το προσωπικό ξέρω ότι είναι σημαντικό να είναι καλά καταρτισμένες οι αντιπροσωπείες, να έχουν προσωπικό δηλαδή που να ξέρει τη δουλειά του καλά. Έχει προετοιμαστεί λοιπόν το προσωπικό των αντιπροσωπιών αυτών για να αναλάβει τέτοια καθήκοντα να μην γίνεται επικάλυψη. Ο κύριος Κουίνς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απαντήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το πρώτο ερώτημα, ποια μέτρα θα λάβει η Ευρωπαϊκή Επίτροπη έτσι ώστε να έχουμε την καλή διαχείριση των προγραμμάτων από τις περιφερειακές οργανώσεις. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιούμε εκτενώς στα περιφερειακά προγράμματα όπου υπογράφουμε ε, συμφωνίες συνεισφοράς, όπως τις αποκαλούμε. Δηλαδή, ε, αντί για χρηματοδότηση ενός συγκεκριμένου προγράμματος, συνεισφέρουμε στον προπολογισμό της οργάνωσης για να συνεισφέρουμε στη δική τους δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας τις δικές τους διαδικασίες, παρά τις δικές μας. Δηλαδή, βασίζονται ε, στα πρότυπα με τις, ε, στα πρότυπα συμφωνιών των Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Τράπεζας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα ταμεία μας, τα κονδύλια, κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και, εν πάση περιπτώσει, η υπογραφή γίνεται μετά από από ε, θεσμικό έλεγχο, έτσι ώστε να δούμε τις διάφορες πτυχές δημοσιονομικής διαχείρισης, όπως τη διαδικασία ε, δημόσιων προμηθειών, ε, εσωτερικούς ελέγχους κλπ. Και με βάση την έκβαση αυτού του ελέγχου μπορούμε να προχωρήσουμε ή όχι. Να υπογράψουμε μία συμφωνία συνεισφοράς. Αυτό και στην Ανατολική και στη Δυτική Αφρική και είχαμε αποκλίνοντα αποτελέσματα. Και μετά, ε, μετά από δύο-τρία χρόνια έχουμε μια έκθεση συνέχειας για να δούμε τι έγινε για να αντιμετωπίσουμε οποιασδήποτε αδυναμίες. Άρα η κομέσα στα πλαίσια των δύο περιφερειών. Η Κομέσα είναι η πιο δυνατή οργάνωση. Είχαμε έναν έλεγχο συνέχειας και στη συμφωνία συνεισφοράς που υπογράψαμε το 2007, η συμφωνία αυτή ε, βαίνει καλός, λειτουργεί καλός. Στην ΣΑΝΤΕΚ που διενεργήθηκε έλεγχος είδαμε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να υπογράψουμε μία συμφωνία συνεισφοράς στα πλαίσια της ΣΑΝΤΕΚ. Και όπως ως προς την ΕΚΟΑΣ και την UMO βρίσκονται κάπου ενδιάμεσα. Έχουμε υπογράψει συμφωνίες αλλά με όρους σε σχέση με τις διαδικασίες δημοσιονομικής διαχείρισης, ιδιαίτερα ως προς τις δημόσιες προμήθειες. Αλλά τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο θετικά, διότι οι οργανώσεις είναι σχετικά αδύναμες. πριν λάβουμε οποιαδήποτε βήματα, διενεργούμε αυτούς τους ελέγχους για να παρακολουθήσουμε την κατάσταση. Σε σχέση με τις αντιπροσωπείες, επειδή είναι περίπλοκο το θέμα των περιφερειών και έχουμε να κάνουμε με πολλαπλότητα περιφερειακών οργανώσεων και πολλές αντιπροσωπείες, θα πρέπει ε, να λάβουμε υπόψη ότι δεν υπάρχει μία ενιαία αντιπροσωπεία που διαχειρίζεται τα περιφερειακά προγράμματα. Και θα μπορούσα να δεχτώ ε, το εξής. Στο παρελθόν δεν συντονίσαμε καλώς τις διάφορες αντιπροσωπείες, προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό και τώρα ζητάμε από τις αντιπροσωπείες στα περιφερειακά προγράμματα να υποβάλουν ε, μία έκθεση σε εξαμηνιαία βάση. Έχουμε επεκτείνει το σύστημα ελέγχου, εξωτερικού ελέγχου προγραμμάτων στο περιφερειακό πρόγραμμα και προσπαθούμε να έχουμε ε, περισσότερο προσωπικό και μπορούμε. Βεβαίως υπάρχει ε, ε, μηδενικός ρυθμός ανάπτυξης, αλλά προσπαθούμε να ενισχύσουμε αυτές τις αντιπροσωπείες κατά το δύνατον. Δεν μπορώ να σχολιάσω την, ε, το 40% απουσίας. Δεν είχα ακούσει στο παρελθόν αυτό το αριθμητικό στοιχείο. Μου φαίνεται υψηλός, ο, υψηλό το ποσοστό απουσίας γιατί σε 12 μήνες το προσωπικό στους 12 μήνες, έχει δύο μήνες άδεια, ε, υπάρχουν και προγράμματα κατάρτισης 10 ε, ημερών και υπάρχουν και αποστολές στα αρχηγεία, σε διάφορα αρχηγεία. Είναι ένα θέμα, αλλά δεν νομίζω ότι φτάνουμε σε ένα 40% σε ένα τόσο υψηλό ε, ποσοστό απουσίας. Αλλά θα πρέπει να το, να το δούμε να δούμε δηλαδή τις αντιπροσωπείες μας και να ενισχύσουμε τις περιφερειακές αντιπροσωπείες εκεί όπου μπορούμε. Σας ευχαριστώ. Εντάχει, γιατί περάσουμε, πρέπει να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Υπάρχει έγγραφο της Κομισιόν για τις αντιπροσωπείες το 2008 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά εγώ έχω κρατήσει και την έκθεση του 2007 και αν θέλετε πολύ ευχαριστώ να σας τα διαβιβάσω. Περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Είναι μια συζήτηση, κοινή συζήτηση που αφορά τα σημεία 5, 6 και 7 της ημερήσιας διάταξης για το, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Γι' αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη δίνω το λόγο στην κυρία Γκρέσλε. Ομιλώ ως εισηγήτρια της Επιτροπής Προϋπολογισμών για το θέμα αυτό, το θέμα δηλαδή του δημοσιονομικού κανονισμού. Εν προκειμένου είμαστε η αρμόδια επιστησία επιτροπή. Θα παρακαλέσω ωστόσο και ε, η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολισμού να αντιληφθεί ότι είναι βασικότατος ο ρόλος της και πρέπει να συμβάλλει. Η Ισπανική Προεδρία σήμερα υποβάλλει συμβιβαστική θέση για την πρόταση την πρόταση Άστον δηλαδή, την οποία έχουμε λάβει επισήμω, αλλά όχι το σχέδιο της Ισπανικής Προεδρία. δηλαδή όχι επισήμω το σχέδιο της Ισπανικής Προεδρίας. Θα κάνω μια πρώτη συνολική αξιολόγηση και της προτάσεω Άστον και της συμβαστική προτάσεω των Ισπανών. Στον τομέα αυτό υπάρχουν τέσσερα δοσιέ. Το πρώτο είναι η ιδρυτική πράξη της ίδιας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας που βρίσκεται στην φάση των ακροάσεων. Δεύτερο, δημοσιονομικός κανονισμός. Εδώ βρισκόμαστε σε πλήρη συναπόφαση. Τρίτο είναι το, το καθεστώς του προσωπικού. Πάλι πλήρη συναπόφαση. Το τέταρτο είναι ο προπολογισμό. Και εδώ βρισκόμαστε στην πλήρη συναπόφαση. Εν, εν αυτού του βαθμού συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναρωτιέται κανείς πώς είναι δυνατόν μέχρι τώρα να μην μας ζητεί κανείς να συνομιλήσουμε. Αυτά που έχουμε λάβει από την κυρία Άστον αποτελούν πρόταση και εγώ νομίζω ότι ως ε, έλεγχος του προϋπολογισμού οφείλουμε να το κρίνουμε προβληματική, υπάρχει ανάμειξη αρμοδιοτήτων. Ανάμειξη αρμοδιοτήτων αντί να είναι ξεκάθαρες. Με βασικό σημείο ότι η εξωτερική υπηρεσία θα ιδρυθεί ως ο οργανισμός εκτός Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αποτέλεσμα να σημειωθούν πολλά νομικά προβλήματα. Και ε, δικαίου της εργασίας του προσωπικού που δεν θα είχαμε εάν η οργάνωση αυτή, η υπηρεσία αυτή αποτελούσε μέρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα μιλήσω για τα προβλήματα αυτά, τα οποία επαναλαμβάνω δεν θα είχαμε εάν εντάσσονταν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα κύριο πρόβλημα είναι η ανάμειξη των αρμοδιοτήτων. Στο μέλλον δηλαδή θα έχουμε έναν επικεφαλής αντιπροσωπείας σε μια τρίτη χώρα, ο οποίος θα διαθέτει χρήματα για όνομα της, στο όνομα της Κομισιόν, χωρίς να είναι μέλος του προσωπικού της Κομισιόν. Μέχρι τώρα αυτό από όψη Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού, αυτό ήταν το λεγόμενο Αγγλιστή no no-go, δηλαδή να μην υπάρχει τέτοια πιθανότητα, να μην υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Άλλωστε και οι ίδιες συνθήκες λένε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτελεί τον προπολογισμό. Μέχρι τώρα ε, τα διάφορα όργανα δεν είχαν παρά έναν επιχειρησιακό προπολογισμό. Όμως υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί που να επιτρέπουν διαχείριση των δαπανών μέσω της εξωτερικής υπηρεσίας. Ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραμένει υπόλογη απέναντί μας. Πόσο ωστόσο θα την καλούμε να είναι υπόλογη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφόσον διαχειρίζουν τα χρήματα άλλοι, εκτός του προσωπικού της. Αυτό λοιπόν θα αποτελέσει σημαντικό πρόβλημα για τον δημοσιονομικό κανονισμό. Γι' αυτό και σε ένα σημείο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει μια νέα πραγματική υπόσταση που είναι η σύγκρουση συμφερόντων. Είναι ενδεχόμενο το οποίο δεν καλυπτόταν μέχρι τώρα νομοθετικά. Και υπάρχουν και special representatives οι οποίοι θα είναι εγκατεστημένοι παρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά δεν θα μπορεί κανείς να ρωτήσει τι κάνουν. Είναι λοιπόν σωστό και σκόπιμο να ζητήσουμε να υπάρξουν ξεκάθαρες αρμοδιότητες εφόσον υπάρχει ένας και μόνο, ένα και μόνο θεσμικό όργανο το οποίο διαχειρίζεται τις δαπάνες, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, βλέποντας το τι πρόκειται να υποβάλει το Συμβούλιο ως συμβαστική πρόταση, συνολικά μπορώ να αξιολογήσω το κείμενο αυτό ότι είναι ακόμα μακρύτερα από τις θέσεις του Κοινοβουλίου. Δηλαδή τα πράγματα που μας ανησυχούσαν έχουν επιδεινωθεί στην πρώτη ανάγνωση του Κορεπέρ. Στο έγγραφο της Ισπανικής Προεδρίας περιλαμβάνονται και οι υπηρεσίες οι οποίες θα υπαχθούν στην υπηρεσία της εξωτερικής δράσεως. Και μέσα στα πλαίσια του Κοινοβουλίου υπάρχει μια steering committee η οποία συμφωνεί ότι θα πρέπει να εγκατασταθεί η Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους κόρπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όντας όμως ένα όργανο sui generis, με μια ιδιαίτερη δηλαδή, νομική βάση, όπως έχουμε περίπου τώρα με την Όλαφ. Εάν γίνει αυτό, θα αποφύγουμε πολλά νομικά προβλήματα. Άλλο πρόβλημα είναι το θέμα του προσωπικού. Από τις χώρες μέλη θα προέλθουν υποτίθεται το 1 τρίτο των ανώτερων αξιωματούχων. Η επιλογή τους όμως είναι θέμα των χωρών μελών. Δεν έχουμε λοιπόν κοινό ορισμό περί του τι σημαίνει διπλωμάτης. η Κομισιόν επιφυλάσσει αυτόν το δικαίωμα να έχει λόγο στο πώς θα επιλεχθούν τα πρόσωπα αυτά. Η Steering Committee, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όλοι οι συντονιστές όλων των επιτροπών, συμφωνεί ότι πρέπει να τεθούν επιτάπητος όλες οι προτάσεις και το καθεστώς του προσωπικού μετά από τις συζητήσεις και με τις επιτροπές προσωπικού θα πρέπει να τεθεί, όπως είπα επιτάπητος, περίπου ε, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Και τέλος είναι και το θέμα του ελέγχου του προπολογισμού. Εμείς θα υποστούμε τις συνέπειες εν τέλει, διότι θα έχουμε να ασχοληθούμε με τις αρνητικές αυτές συνέπειες χρόνο με το χρόνο. Και δεν θα υπάρχουν και καθαρά υπόλογοι απέναντί μας. Σας ευχαριστώ κύριε Γκρέσλη. Το λόγο έχει ο ο κύριος Κάλφιν για ένα άλλο θέμα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να συμμετάσχω και εγώ στην προκαταρτική αυτή συζήτηση, στηρίζοντας πολλά από τα σχόλια της κυρίας Γκρέσλερ. Και θα προσπαθήσω να πάω και ακόμα πιο μακριά. Είναι πολύ βασικό να λάβουμε υπόψη μας νέα προβλήματα που δημιουργούνται όσον αφορά τις δημοσιονομικές διαδικασίες από τη δημιουργία ενός νέου οργάνου. Όπως ήδη είπε η κυρία Γκρέσλερ, δεν έχουμε ήδη υπάρχοντες μηχανισμούς που να μας επιτρέπουν με σωστό τρόπο να σχεδιάζουμε, να εφαρμόζουμε και να ελέγχουμε και να χρησιμοποιούμε χρήματα από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους. Η μία λύση που έχουμε είναι να προσπαθήσουμε να κολλήσουμε την υπηρεσία εξωτερικής δράσης σε έναν από τους ήδη υπάρχοντες μηχανισμούς. Αυτό είπε και η κυρία Κρέσελ και αυτό υπάρχει και στο non-paper, την πρόταση που έχουμε από τον κύριο Μπρόκεφ Χώστατ. Κατά τη γνώμη μου αυτή θα είναι μια πολύ καλή λύση αν περάσει στο Συμβούλιο. Όμως πιστεύω ότι θα υπάρξει αντίσταση από πλευράς του Συμβουλίου σε μια τέτοια λύση. Αν λοιπόν δεν χρησιμοποιήσει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης τους μηχανισμούς που ήδη ισχύουν για άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο μηχανισμό, τον οποίο πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ καλά, για να λειτουργήσει ο νέος αυτός θεσμός. Όταν μιλάμε για μια προσέγγιση όσον αφορά ένα νέο όργανο, εμείς στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού, πρέπει να δούμε κατά πόσο εφαρμόζονται διάφορες αρχές, όπως είναι η υπευθυνότητα, η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα, η απόδοση. Το βασικό πρόβλημα, λοιπόν, το κύριο πρόβλημα το οποίο δημιουργείται σε περιπτώσεις όπως αυτή η Generis υπηρεσία εξωτερικής δράσης, προέρχεται από το γεγονός ότι θα είναι δύσκολο να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Έχουμε διάφορα έγγραφα και αυτά που προτείνει η ίδια Καθνάστον και έγγραφα από ευρωβουλευτές κλπ. κλπ. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής διάκριση στις αρμοδιότητες των δύο οργάνων. Και φοβάμαι ότι ό,τι και αν κάνουμε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα είναι σε θέση να δημιουργήσει με σαφήνεια μια ξεκάθαρη εικόνα διακριτών αρμοδιοτήτων ανάμεσα στα δύο όργανα. Και εκείνοι που ερχόμαστε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στα στοιχεία εκείνα απαλλαγή σε δύο επίπεδα. Πρώτον, συντονισμός ανάμεσα στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως λένε και πολλά γραφά, θα υπάρχει οριζόντια κατανομή αρμοδιοτήτων. Ο σχεδιασμός θα γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διορθώνει ο μιλητής. Ο σχεδιασμός θα γίνεται από την εξωτερική δράση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ασχολείται με τη χρήση των κονδυλίων. Λυπούμε λοιπόν, γιατί όταν προσπαθώ να δω αυτή την αλυσίδα αρμοδιοτήτων που συνδέει το σχεδιασμό με την χρήση των κονδυλίων, διαπιστώνω ότι θα αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά προβλήματα εξαιτία της ασάφειας αυτής όσον αφορά τις αρμοδιότητες των δύο οργάνων. Άρα πρέπει να επικεντρωθούμε στους μηχανισμούς συντονισμού, συμπεριλαμβάνοντας πρωτοβιουλίες, τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις, συμπεριλαμβάνοντας την ε, παρουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πώς θα εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τέλος βέβαια σχεδιασμός και ε, χρήση των κονδυλίων. Το δεύτερο επίπεδο συντονισμού πρέπει να γίνεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εδώ είναι ένα θέμα που ίσως δεν έχει άμεσα σχέση με την εγκαθίδρυση της Υπηρεσία εξωτερικής δράσης, αλλά όταν μιλάμε για την αναδιάρθρωση του προπολογισμού, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το συντονισμό μεταξύ του ε, Πρόεδρου της Επιτροπής και των τριών Επιτρόπων. Πρώτον, λοιπόν, περισσότεροι προσοχή στις λεπτομέρειες όσον αφορά το συντονισμό, όσον αφορά τις αρμοδιότητες των διαφόρων οργάνων. Δεύτερον, ποιος λογοδοτεί, πώς. Φυσικά και υπάρχει υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες που έρχεται και λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το σώμα, αλλά και όσον αφορά τον προπολογισμό. Εδώ τα ερωτήματα είναι πολλά. Εξάλλου και στο έγγραφο των κύριων Μπροκ και Φερχόσταφ, έχουμε εδώ μια τελευταία εκδοχή. Υπάρχουν πολλές καλές ιδέες και κάποιες εναλλακτικέ λύσεις. Πρέπει να βασιστούμε σε πολλοί κέρες αρχές. Πρώτον, εκπροσώπησε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ποια είναι η θέση των αναπληρωτών της ΥΠΑ του. Δύο αναλλακτικέ λύσεις προτείνονται από τους συναδέρφους ή ορίζονται με πρωτοβουλία του Συμβουλίου ή προτείνονται από την ύπατο εκπρόσωπο με ειδική πλειοψηφία ε, ψηφίζει το Συμβούλιο στη συνέχεια. Προτιμώ τη δεύτερη επιλογή για να υπάρχει ισορροπία. Αλλιώ είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρουμε ποιο είναι υπεύθυνο γιατί, για ποιο πράγμα. Πρέπει να ξέρουμε ότι η τελική ευθύνη για μερικά πράγματα την έχει η ύπατο εκπρόσωπο και για άλλα ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όταν ε, λέμε ποιο λογοδοτεί και πώ, εδώ έχουμε να κάνουμε και με τους μηχανισμούς ε, ορισμού και με τον έλεγχο. Είπε και η κυρία Γκρέσλερ ότι είναι δύσκολο γιατί η διαδικασία μας τι λέει, είπαμε, το σχεδιασμό τον κάνει η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την εφαρμογή και τη χρήση των κονδυλίων την Επιτροπή. Μετά πάμε πίσω στην Υπηρεσία Εξωτερικών, ε, Εξωτερικής Δράσης Είναι δηλαδή μια, ένα πινκ-πονγκ ευθύνη που πηγαίνει από τον ένα στον άλλον και που θα δημιουργήσει προβλήματα. Όταν λοιπόν μιλάμε για τους ορισμούς και τις αρμοδιότητες των ε, υψηλά εισταμένων και στην Επιτροπή και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Έπειτα, για τα δημοσιονομικά που είναι και αυτό που ενδιαφέρει την Επιτροπή μας. Στην πράξη τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι θα χωρίσουμε τον προπολογισμό που είναι για την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που σήμερα είναι στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή και θα μετατοπιστεί και θα πάει στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή πρέπει να διαχωριστούν οι διοικητικέ δαπάνες και να δημιουργήσουν μια διαδικασία απαλλαγή για την εξωτερική δράση όσον αφορά τις διοικητικέ δαπάνες. Γι' αυτό πρέπει να τροποποιηθεί ο δημοσιονομικός κανονισμός για να γίνει αυτό. Πάντως, ο διαχωρισμός των ε, δαπανών σε διοικητικές και λειτουργικές θα είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Από όσο ξέρω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχει ζητήσει πολλές φορές να έχει πληροφορίες, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, όσον αφορά την διάκριση των διοικητικών και λειτουργικών δαπανών και δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Το καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολο να γίνει ο διαχωρισμός αυτός. Οπότε μένει το ερώτημα ποιος θα είναι υπεύθυνο γιατί και κατά πόσο οι διοικητικές δαπάνες που θα είναι της ε, εξωτερικής δράσης θα καλύπτει όλες τις διοικητικές δαπάνες ή τις δαπάνες που θα έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα υπάρχουν κάποιες επιπλέον δαπάνες για τη δίκηση. Πρέπει να σκεφτούμε μήπως σαν ενημέρωση να έχουμε έναν παγιωμένο προπολογισμό που να περιλαμβάνει και τον προπολογισμό της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης και τα κονδύλια τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στην εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό για να έχουμε μια ιδέα των συνολικών δαπανών που πάνε στις εξωτερικές μας δράσεις. Δεν νομίζω ότι έτσι καλώς μπορούμε να αλλάξουμε τις δημοσιονομικές διαδικασίες, αλλά αυτή την πληροφορία μπορούμε κάλλιστα να τη ζητήσουμε. Το συνολικό δηλαδή προπολογισμό, ώστε να ξέρουμε συνολικά τι κονδύλια πηγαίνουν στην εξωτερική μας δράση. Και ολοκληρώνω με δύο προβλήματα. Τα αναφέρω απλώς. Το θέμα της επικάλυψης και το θέμα του ουδέτερου προπολογισμού της νέας υπηρεσίας. Όταν μιλάμε για επικάλυψη, το Κοινοβούλιο έχει πει μέχρι τώρα ότι δεν πρέπει να υπάρχουν επικαλύψεις. Και να μην υπάρξουν νέα επιπλέον δαπάνες για την υπηρεσία, να μην επηρεαστεί ο προπολογισμό. Όμως στην πράξη είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί αυτό. Η μεταφορά προσωπικού από το Συμβούλιο και την Επιτροπή προς την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει αύξηση στον προπολογισμό, αλλά κάποιες μονάδες πρέπει να παραμείνουν και ο διοικητικός ε, προϋπολογισμός, τα διοικητικά κονδύλια δεν θα είναι ακριβώς τα ίδια στην Επιτροπή, το Συμβούλιο και την ε, νέα υπηρεσία, άσε που θα έρθουν και διπλωμάτες από τα κράτη-μέλη. Και αυτό θα επιβαρύνει βέβαια τον προπολογισμό. Και το άλλο το οποίο κάλυψε βέβαια βρέως η κυρία Γκρέσλερ είναι το θέμα της επικάλυψης. Προτείνει να είναι επιτροπή να φροντίζει για τη για τον τρόπο που θα λειτουργεί η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να αφαιρέσουμε από την υπηρεσία εξωτερικής δράσης την δυνατότητα η ίδια να κανονίζει τις διοικητικές της δαπάνες. Έτσι κινδυνεύουμε να βρεθούμε με επικαλύψεις που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσπαθήσει να περιορίσει όσο γίνεται περισσότερο. Αυτά είναι τα κυρία ζητήματα που έχω εντοπίσει εγώ. Ευχαριστώ. Σε σχέση με την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου για το σημείο 2 δίνω το λόγο στον κύριο Ριβελίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σήμερα συζητάμε την πρόταση κανονισμού του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό του 2002 για τον Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δυνάμει του κανονισμού 1605 κάθετος 2002. Επειδή υπάρχουν ε, συνάδελφοι που δεν παρακολούθησαν το θέμα, θα ήθελα να σας μιλήσω για το, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Και για αυτή την υπηρεσία έχουμε τέσσερις διαφορετικές πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, αλλά έχουν αποδοθεί οι πρώτες δύο πράξεις. Η, πράξεις. η πρώτη είναι μία νομοθετική πράξη του Συμβουλίου για τη λειτουργία της υπηρεσίας απόφαση του Συμβουλίου όπου έγινε ε, διαβούλευση με το ε, άφετ, με την ΑΦΕΤ μόνο. Η δεύτερη είναι μια πρόταση τροποποίησης του δημοσιονομικού κανονισμού, ε, τακτική νομοθετική διαδικασία σε συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και ο υποφαινόμενος είναι εισηγητής. Η τρίτη είναι μια πρόταση πρόταση για να αλλάξουμε το καθεστώς του προσωπικού Γιούρι Βασική Επιτροπή και η συγγετής είναι ο συνάδελφος Χέρτζοκ, τέταρτη πράξη, τροποποιητικός κανονισμός για το 2010 και ε, η συγγετής είναι ο κύριος Μπαλτσίτης. Από τις ε, τέσσερις προτάσεις, δύο έγιναν αποδεκτές από το Κοινοβούλιο. Η πρώτη πρόταση που σας ανέφερα και ο δημοσιονομικός κανονισμός, δηλαδή η δεύτερη πρόταση, όπου εγώ είμαι εισηγητής. Και θα ήθελα να ζητήσω από τον εκπρόσωπο της Επιτροπής να μου πει πότε πιστεύετε ότι αυτές οι προτάσεις θα φτάσουν επιτάπητος, διότι θα πρέπει να προβούμε σε μια επιλογή για να μην πρέπει να αποφανθούμε και για τις τέσσερις. Η πρώτη τροποποίηση του Δημοσιονομικού Κανονισμού υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 24 Μαρτίου 2010 μαζί με ένα έγγραφο εργασίας για τις τροποποίησεις που απαιτούνται για τον τρόπο εκτέλεσης του Δημοσιονομικού Κανονισμού σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Επί της πρότασης αυτής θα ασχοληθώ με θέματα αποκλειστικά της δικής μου αρμοδιότητας, αν και είναι δύσκολο να ορίσουμε ένα γενικό πλαίσιο χωρίς να λάβουμε υπόψη τις θέσεις των άλλων επιτροπών επί του θέματος. Όπως είπαμε, στην πρόταση του Συμβουλίου η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης είναι μια υπηρεσία, αυτόνομη υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεχωριστή από την Κομισιόν και από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου. Υπό την ε, ύπατη εκπρόσωπο και θεωρείται θεσμικό όργανο καθε αυτό. Θα έχει μια κεντρική διοίκηση και αντιπροσωπείες ε, σε όλο τον κόσμο θα βοηθήσει στο έργο της ΥΠΑ της εκπροσώπου για τις εξωτερικές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα καλύπτουμε όλες τις χώρες του κόσμου και ειδική θεματική, ειδικές θεματικές για τις ε, ε, πολύπλευρες σχέσεις. Μπορούμε να επικρίνουμε όμως μερικές πτυχές του έργου. Σύμφωνα με την ε, έκθεση, ο φορέας που θα είναι υπεύθυνο για, το, για θέματα διοικητικού φόρτου και υπεύθυνο για τις απαλλαγές δεν αλλάζει το άρθρο 145 του Δημοσιονομικού Κανονισμού που ορίζει τους κανόνες περί απαλλαγής. Η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει ότι ο δικαιούχος της απαλλαγής, δυνάμει του άρθρου 319, ο δικαιούχος είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα, έχει, δεν θα μπορέσει να επηρεάσει την κατάσταση τη στιγμή που ο δικαιούχος της απαλλαγής δυνάμει του άρθρου 319 είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το, η δεύτερη επίκριση είναι ότι η παρούσα πρόταση της ΥΠΑ ε, ΕΕ της εκπροσώπου της ε, Επιτρόπου Άστον ορίζει ότι θα υπάρχουν επιπτώσεις πολύ σημαντικές και ούτε ο πρόεδρος Μπούζεκ δεν θα μπορέσει να επηρεάζει τη διαδικασία. Τρίτο σημείο κριτικής. Ο εισηγητής της Επιτροπής ΑΦΚΟ, κ. Φερχόφστατ, υπογράμμισε ο ίδιος το εξή ότι η συνθήκη δεν ε, κάνει μνήα του νέου οργάνου και δεν θεωρεί ότι πρόκειται για νέο οργανισμό. Κατά συνέπεια, πρέπει να συνδεθεί με ένα άλλο όργανο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ας πούμε. Ο συνάδελφος Φερχόφστατ και εγώ δεν ερχόμαστε από το ίδιο κόμμα, αλλά επί αυτού συμφωνούμε. Συνεχίζω λοιπόν αναλύοντας την πρόταση και διαπιστώνω ότι σύμφωνα με την πρόταση αυτή η καθημερινή διαχείριση της υπηρεσίας θα είναι αρμοδιότητα ενό γενικού γραμματέα με, δύο με έναν αναπληρωματή και δύο βοηθού, και διαπιστώνω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για το Ταμείο ανάπτυξη, του Ευρωπαϊκού Οργάνου για τη Δημοκρατία κλπ. κλπ αλλά θα συνεργάζεται στενά με τον, την εκπρόσωπο, την είπα, το εκπρόσωπο και τις υπηρεσίες. Ε, όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως, κατά τη σύνταξη της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο, ο διαχωρισμός εργασίας θα είχε ως εξής. Ο, η υπηρεσία θα είναι υπεύθυνη για τις στρατηγικές αποφάσεις, στρατηγικά έγγραφα για τις περιφέρειες και τις χώρες και εθνικά ενδεικτικά προγράμματα, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση όλων αυτών των προγραμμάτων. Όμως θα πρέπει να διευκρινίσουμε ε, κάτι το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια σύγχυση, η οποία δεν είναι ηθελημένη ορισμένες ε, τροποποίησεις του άρθρου 49 του Δημοσιονομικού Κανονισμού που αφορούν ε, τις βασικές νομοθετικές πράξεις δυνάμει του τίτλου 5 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης υπάρχουν μόνο στην πρόταση τροποποίησης για την, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στη συνθήκη της Λισαβόνας. Αλλά δεν υπάρχουν σε αυτή την πρόταση. Νομίζω ότι αυτές οι προβλέψεις θα πρέπει να αναλυθούν εν λεπτομερία και θα ήταν σκόπιμο να ε, το κοινοποιήσουμε και στην νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να διευκρινιστεί είναι αυτό που σχετίζεται με τις αντιπροσωπίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο. Υπεύθυνοι θα είναι οι επικεφαλής αντιπροσωπείων ε, που θα διοριστούν από την ύπατη εκπρόσωπο. Στους τομείς λοιπόν που υπάρχει αρμοδιότητα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι επικεφαλής θα λαμβάνουν οδηγίες και από την Κομισιόν. Στην πρόταση λέμε στην ουσία ότι οι επικεφαλείς αντιπροσωπιών επειδή είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του προϋπολογισμού θα είναι υπόλογοι ενώπιον των γενικών διευθυντών και τελικά ενώπιον της Επιτροπής. Η πρόταση δεν διευκρινίζει την κατανομή αρμοδιοτήτων και την γεωγραφική, θα μπορούσα να πω, κατανομή αρμοδιοτήτων το ζήτημα οδηγεί σε σύγχυση για τις ορισμένες μεταφράσεις, ιδιαίτερα στα αγγλικά, ιταλικά και γερμανικά. Το άρθρο 50 του Δημοσιονομικού Κανονισμού θα οδηγούσε σε αμφιβολίες σε σχέση με ορισμένα λειτουργικά έξοδα του προϋπολογισμού. Εάν η διατύπωση δεν αλλάξει, τότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ορισμένες δαπάνε που θα ορίζει η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να τροποποιήσουμε την πλαισίωση αυτή για να μην υπάρχει σύγχυση. Τέλος, η πρόταση δεν μιλά για τον αριθμό ε, διπλωματών από την Επιτροπή, Κοινοβούλιο και Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου. Αναφέρουμε μόνο ότι θα λειτουργήσει πλήρως η υπηρεσία με εν τρίτον του προσωπικού που θα προέρχεται από διπλωμάτες των κρατών μελών. Και ο πρόεδρος Μπούζεκ τόνισε ότι στη διαδικασία startup θα πρέπει να συμμετέχουν και οι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει να έχουμε έναν τουλάχιστον ε, υψηλό βαθμό υπάλληλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ως προς το προσωπικό και πάλι ως προς το προσωπικό φαίνεται ότι σε επίπεδο κορεπέρ ορισμένα κράτη-μέλη τόνισαν ότι θα ήθελαν να είναι αρμόδια για το προσωπικό, αποκλειστικά δηλαδή τα κράτη-μέλη, ε, και να είναι υπόλογα στην κυρία Άστον ή στη Γενική Γραμματεία. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι είπαν και οι τρεις εκπρόσωποι των βασικών πολιτικών ομάδων όπου μίλησαν για ένα διακυβερνητικό πρότυπο, το οποίο θα πρέπει να ισχύσει. Ένα άλλο βασικό ζήτημα αφορά την πρικοδότηση. Ακόμα δεν έχουμε αριθμητικά στοιχεία, συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Έχουμε μόνο φήμες και αντικρουόμενες. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή κατά πόσο μπορεί να μας δώσει αυτά τα αριθμητικά στοιχεία. Πόσα θα δαπανίσετε για τις αντιπροσωπείες της, ε, και πόσα δαπανάτε για τις αντιπροσωπείες της Κομισιόν ανά τον κόσμο και πόσο θα δαπανίσετε στο μέλλον. Ε, θα υπάρχει άμεσος έλεγχος μέσα στα πλαίσια της υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Τέλος, όσα αφορά τους επικεφαλείς αντιπροσωπιών, τίποτα δεν ελέγχθη ως προς τη δυνατότητα να γίνονται ακροάσεις πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Θα ήθελα η Επιτροπή και το Συμβούλιο να μου διευκρινίσει αυτό το σημείο. Τέλος, στο πρώτο σημείο, έχοντας λάβει υπόψη την δημοσιονομική οργάνωση του οργανισμού, επειδή πρόκειται για αυτόνομο οργανισμό και επειδή δεν εντάσσεται στον ε, μηχανισμό απαλλαγής στρίκτο σένσου του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να υπάρξει αυτός ο διαχωρισμός. Και επειδή ε, δεν υπάρχει διασάφηση του δημοσιονομικού καθεστώτος, σε σχέση με τους επικεφαλείς αντιπροσωπιών θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε αυτό το σημείο. Τρίτον, λαμβάνοντας υπόψη της τροποποίησης του άρθρου 50 για ορισμένα λειτουργικά έξοδα δημοσιονομικού ελέγχου θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Επειδή μέχρι σήμερα δεν υπάρχει πρόταση επάνδρωσης του προσωπικού, θα πρέπει να έχουμε μελλοντικά στοιχεία και θα πρέπει να υπάρχει ε, διαχωρισμός διοικητικών και λειτουργικών εξόδων. Γι' αυτό δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη η παρούσα πρόταση. Λαμβάνοντας τις τροποποιήσεις του άρθρου 44, δυνάμει της νέας συνθήκης της Λισαβόνας, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς τη διαχείριση να λάβουμε υπόψη το ψήφισμα της 22ης ε, Οκτωβρίου 2009 ως προς την δημιουργία Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και επειδή σήμερα δεν υπάρχουν σαφή αριθμητικά στοιχεία για την πρικοδότηση του φορέα αυτού, νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει όλες τις προτάσεις που εντάσσονται στην αξιολόγηση αυτού του κανονισμού, στο σύνολό τους. Άρα θα ήταν ευκταίο να, έχουμε, να κάνουμε με μια αυτόνομη υπηρεσία, η οποία όμως να ενσωματώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι αυτό το πρότυπο είναι το καλύτερο ως προς τη δημοσιονομική διαχείριση και επάνδρωση προσωπικού. Άρα θα ήταν σκόπιμο να προβούμε στην εκείνη αναθεώρηση του δημοσιονομικού πακέτου, δηλαδή μια παράλληλη αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να προσαρμοστούμε στη συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Επειδή δεν έχουμε μία πλήρη ε, πλαισίωση, δεν μπορώ να γνωμοδοτήσω θετικά στην πρόταση. Και κάνοντας και μία πολιτική αξιολόγηση, θα ήθελα να πω τα εξής. Είναι σαφές ότι το Συμβούλιο ε, επειδή στο Συμβούλιο συμμετέχουν ε, ε, χώρες που χρηματοδοτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος και βεβαίως η Επιτροπή βρίσκεται σε μια φάση αναποφασιστικότητας. Αλλά στα πλαίσια του δημοκρατικού ελέγχου που γίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να υλοποιήσει αυτό τον έλεγχο. Και δεν μπορούν να του αφαιρεθούν οι αρμοδιότητες στα πλαίσια της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Ευχαριστούμε. Σε σχέση με την ε, τρίτη πρόταση έχουμε τον κύριο Χέρτσοκ, τον οποίο δεν βλέπω. Και άρα περνάμε στον κύριο Μπάλτσιντης. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι τρεις που πήραν το λόγο πριν από μένα εντόπισαν διάφορα προβλήματα. Και πράγματι υπάρχει το ζήτημα. Η δημιουργία αυτής της υπηρεσίας επιλέχθηκε ως η πιο περίπλοκη εναλλακτική. Στον προπλησμό του 2010 υπάρχουν ε, τροποποίησεις, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια νέα δομή. Μια νέα δομή θα προβλεφθεί όταν ληφθούν αποφάσεις για τροποποίησεις των δημοσιονομικών κανονισμών και κανονισμών όσον αφορά το προσωπικό. Εμείς οι τέσσερις λοιπόν συντάκτες γνωμοδοτήσεων συζητάμε μεταξύ μα Και βάσει των πληροφοριών που έχουμε μέχρι τώρα, η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του προπολογισμού 2010 θα υποβληθεί τον Ιούνιο. Τότε θα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα και για μας. Τώρα μιλάμε για αμφιβολίες, για παρατηρήσεις που έκαναν και οι προλαλήσαντες, που υποστηρίζω απόλυτα κι εγώ. Το Κοινοβούλιο που προχώρησε με τη νέα Επιτροπή Μπαρόσο τώρα αντιμετωπίζει την δημιουργία ενός νέου οργάνου, το οποίο δεν ελέγχει καθόλου. Συμφωνώ με την κυρία Κρέσλερ πάντως ότι και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνεργάζονται πολύ περισσότερο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πιο στενά. Σε ένα χρόνο θα αξιολογήσουμε τις δραστηριότητες του νέου οργάνου και την ε, απόδοση λογαριασμών. Πώς έχουν χρησιμοποιήσει τα κονδύλια που τους έχουμε διαθέσει. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν πρώτα να λυθούν τα σοβαρά προβλήματα που εντόπισαν οι συνάδελφοί που πήραν το λόγο πριν από μένα και μόνο τότε να μιλήσουμε για νέα κονδύλια όσον αφορά τη λειτουργία αυτής της υπηρεσίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στη συνέχεια. Στα μέλη της Επιτροπής θα ήθελα να πω ότι και προσωπικά συμμετείχα με την κυρία Γκρέσλε στην ε, ομάδα της Ευρωπαϊκή, του Ευρωπαϊκού Συνοβουλίου υπό τον ε, πρόεδρο κύριο Μπούζεκ και θίξαμε ε, ορισμένα Σημεία δηλαδή ότι η Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και να μην επικαλύπτεται από άλλους, διότι πρόκειται για πολύ σημαντικά θέματα για το πώς δαπανώνται τα ε, χρήματα της υπηρεσίας αυτής. πρέπει να λάβουμε υπόψη και μία σειρά δαπανών που δεν έχουν οριστεί. Βεβαίως και το θέμα του προσωπικού είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα δεν υπάρχει σαφήνεια. Ήδη στο παρελθόν ανέκυψαν προβλήματα στο, σε τομείς συνεργασίας όπου συμμετέχει και η ύπατη εκπρόσωπος ιδιαίτερα σε περιοχές, σε τομείς όπου υπάρχει ε, ρήξη συμφερόντων. Αύριο θα σας πω τι συμβαίνει και με το θέμα του Αφγανιστάν, διότι μας ενδιαφέρουν και οι ζώνες σύραξης. Άρα θα πρέπει και ο πρόεδρος Μπούζεκ να παρέμβει έτσι ώστε η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον ε, έλεγχο αυτής της υπηρεσίας και στα πλαίσια της Επιτροπής και ως ε, ανεξάρτητος οργανισμός. Αυτό ανέκυψε και από την παρούσα συζήτηση, δηλαδή τον κεντρικό ρόλο της δικής μας Επιτροπής. Και θα δούμε τι θα ανακύψει από την Επιτροπή και από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου. Ο κύριος Γουανγιέν έχει το λόγο. Euh, Ευχαριστώ. Άκουσα πολύ προσεκτικά όλα όσα είπαν οι εισηγητές σας. Πριν μπω στην ουσία, όμως, επιτρέψτε μου να δώσω κάποιες διευκρινήσεις για το χρονοδιάγραμμα, μια που και αυτό αναφέρθηκε όπως συμφωνήθηκε. Πήρατε τις προτάσεις της κυρίας Άστον για το σχέδιο απόφασης. Είναι μια επίσημη θέση. Έχετε και την πρόταση τροποποίησης του δημοσιονομικού κανονισμού, αλλά δεν έχετε ακόμα την επίσημη πρόταση τροποποίησης του καταστατικού. Και αυτό για τον απλούστατο λόγο ότι, ότι πρέπει να τηρηθούν κάποιες διαδικασίες, δηλαδή να υπάρξει πρώτα διαβούλευση με τα συνδικαλιστικά όργανα. Μόνο αφού έχει γίνει η διαβούλευση με τα συνδικαλιστικά όργανα, με τους εκπροσώπους δηλαδή τον του προσωπικού, μόνο τότε η Επιτροπή θα είναι σε θέση επίσημα να υποβάλει την πρότασή της. Δεν πρόκειται για καθυστέρηση, αλλά πρόκειται για μια διαδικασία η οποία παίρνει λίγο παραπάνω χρόνο παραπάνω από όσο η τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Τώρα για τον διορθωτικό προπολογισμό. Η πρόταση αυτή θα υποβληθεί, το έχω πει κι αλλού, εξάλλου, όσο γίνεται πιο γρήγορα. Σε εσωτερικό επίπεδο προχωράμε πολύ καλά σχετικά με τον ορισμό του προσωπικού που θα αποσπαστεί είτε από το Συμβούλιο είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την αυτή Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να προχωράμε γρήγορα. Θα ολοκληρώσουμε το σχέδιο του ιδιωτικού προϋπολογισμού, όπως και να έχει το πράγμα, από τη στιγμή που έχουμε όλα τα οριστικά, τα τελικά δεδομένα. Μετά θα γίνει μια εσωτερική δουλειά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα κρατήσει τέσσερις περίπου εβδομάδες. Κατόπιν τούτων, Πρόεδρε, θέλω να επανέλθω στην ουσία. Σε αυτά που είπαν οι διάφοροι συγητές. Υπάρχει μια επιλογή που γίνεται Την κάνουν οι ομάδες οι οποίες σχεδιάζουν την ανάπτυξη της υπηρεσίας αυτής. Και η επιλογή αυτή είναι να έχει μία κάποια αυτονομία αυτή η υπηρεσία. Είναι μια υπηρεσία η οποία δημιουργήθηκε από τη συνθήκη υπό την ευθύνη της ε, είπα του εκπροσώπου και η επιλογή έγινε σε πολιτικό επίπεδο να υπάρχει αυτή η αυτονομία. Να δώσουμε δηλαδή ένα βαθμό ανεξαρτησίας. Αρκετά μεγάλο στην υπηρεσία αυτή, παρόλο που η ίδια συνθήκη δεν λέει ότι πρόκειται για ξεχωριστό θεσμικό όργανο. Δημοσιονομικά τώρα αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι μας ζητήθηκε να φτιάξουμε την υπηρεσία περίπου όπως θα φτιάχναμε ένα καινούριο όργανο. Αυτό δημοσιονομικά σημαίνει ότι η υπηρεσία αυτή πρέπει να έχει στη διάθεσή της και δημοσιονομική αυτονομία όσον αφορά τις διοικητικές της δαπάνες. Δεδομένου ότι ο λειτουργικός προϋπολογισμός της εξακολουθεί να παραμένει στα χέρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκείνη ελέγχει. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό είναι ένα στοιχείο κλειδί στην ε, προσέγγιση της. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν λειτουργικές δαπάνες να φεύγουν από τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήταν αντίθετο και στη συνθήκη στο κατά αυτό. Εμείς λοιπόν καλούμεθα να ελέγξουμε ότι τηρείται αυτό και να φροντίσουμε ότι παρόλα αυτά η εξωτερική αυτή η δράση, η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα δρά αποτελεσματικά και από πλευράς προπολογισμού. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε είναι εκείνο της έλλειψης συνέχειας. Δηλαδή, από τη μια στιγμή έχουμε την, από μια μεριά έχουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την άλλη μεριά έχουμε τους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών. Εκεί λείπει ένας κρίκος. Η Κομισιόν διαχειρίζεται είτε από την έδρα της, είτε αποκεντρωμένα μέσω των διαφόρων αντιπροσωπιών τα διάφορα κονδύλια. Οι επικεφαλής των αντιπροσωπιών έχουν όντως κάποια ε, δημοσιονομική ευθύνη. Στο σχήμα που έχουμε εμείς σήμερα στα χέρια μας, οι επικεφαλείς των αντιπροσωπιών δεν είναι πια ε, υπάλληλοι της Κομισιόν και άρα δεν μπορούν πια να ασκήσουν τον ίδιο ρόλο όπως είχαν πριν δημιουργηθεί η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Συγχρόνως, εμείς που θέλουμε μια αποτελεσματική υπηρεσία βέβαια, αναρωτηθήκαμε πώς μπορεί αυτό να διακανονιστεί εξακολουθώντας να έχουμε υψηλής ποιότητας ελέγχους. Προχωρήσαμε προς την κατεύθυνση που λέει ότι πρέπει λίγο πολύ να ξαναφτιάξουμε τη σύνδεση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών. Να αποκατασταθεί δηλαδή αυτή η αλυσίδα, αυτή η σχέση κάθε επικεφαλής αντιπροσωπείας με την Επιτροπή, έτσι ώστε η Επιτροπή να ξέρει ότι οι κανόνες όσον αφορά την χρηστή διαχείριση τηρούνται. Προβλέψαμε για να μπορέσουν οι υποκεφαλείς των αντιπροσωπείων να μπορούν να λειτουργήσουν ως πρέσβεις εντός αγωγικών και να μπορούν να εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στο δημοσιονομικό, ήταν σημαντικό να μπορούν να συνεχίζουν να έχουν τις αρμοδιότητες που είχαν μέχρι την δημιουργία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Βέβαια, η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι η Επιτροπή έχει και αυτή λόγο για την επιλογή του επικεφαλής αντιπροσωπείας. Είναι πολύ βασικό αυτό για την Κομισιόν. Και δεύτερον, στα πλαίσια της ε, βοήθειας που θα ζητάμε, οι υποδιατάκτες εξακολουθούν να είναι υπεύθυνοι για όλες τις δημοσιονομικές λειτουργίες θα τηρούν τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν να κάνουν με την εκτέλεση του προπολογισμού βάσει των ίδιων υποχρεώσεων και δικαιωμάτων όπως και όταν ε, εκπροσωπούσαν την Επιτροπή. Και οι ίδιες οδηγίες θα δίνονται στους επικεφαλείς των αντιπροσωπιών. Οι κανόνες θα εξακολουθούν να εφαρμόζονται και να ισχύουν και ειδικό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει να κάνει με ατασταλείς θα είναι υπεύθυνο για να παρακολουθεί τις περιπτώσεις εκείνες που μπορεί να προκύψουν. Συνεπώς, επ' αυτού νομίζω ότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Θα παραμείνουμε μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγχει πλήρως τις δαπάνες που θα συνεχίσουν, τις λειτουργικές δαπάνες που θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται οι αντιπροσωπείες, γνωρίζοντας όμως ότι στην κάθε αντιπροσωπεία θα υπάρχει στήριξη από τις μονάδες συνεργασίας που θα ελέγχονται από τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, ξαναφτιάξαμε αυτή την αλυσίδα που μας επιτρέπει να διατηρήσουμε ένα επίπεδο τουλάχιστον ίδιο όσον αφορά την ποιότητα διαχείρισης των οικονομικών. Επιτρέψτε με εδώ τώρα να κάνω και μια δεύτερη παρατήρηση. Σχετικά με πιο συγκεκριμένα τα κονδύλια της ε, εξωτερικής ε, πολιτικής. Όλα αυτά τα κονδύλια τα διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το συζητάνε σήμερα οι Υπουργοί, αλλά ζητήσαμε ότι οι ομάδες οι οποίες διαχειρίζονται αυτά τα κονδύλια να εξακολουθούν να βρίσκονται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ακόμα κι αν είναι απόλυτα εφικτό, την ευθύνη τους να την έχει η ύπατος εκπρόσωπος ως όμως αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα είναι υπάλληλοι αυτοί οι οποίοι δεν θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Τουλάχιστον σήμερα αυτή είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιμένει σε αυτήν. Έρχομαι τώρα στο σχεδιασμό. Εδώ πάλι πρέπει να διευκρινίσουμε τα πράγματα. Η σύλληψη του σχεδιασμού, για να είμαστε πολιτικά συνεπείς, εξασφαλίζεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, πράγματι. Αλλά οι αποφάσεις που έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό και οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση είναι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως σώμα, συλλογικά. Δεν υπάρχει δηλαδή διαφορά σε σχέση με την σημερινή διαδικασία. Τέλος, πρόεδρε, ακόμα και αν υπάρχουν ακόμα πολλά σημεία που θα ήθελα να σχολιάσω, αλλά φαντάζομαι ότι ο χρόνος πιέζει, θέλω να πω δύο λόγια ακόμα για το θέμα της λογοδοσίας. Στο βαθμό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να είναι υπεύθυνη για την διαχείριση όλων των λειτουργικών δαπανών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να είναι υπόλογος για όλες τις δράσεις που αναπτύσσονται σε αυτά τα πλαίσια. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η κυρία Άστον είχε την ευκαιρία να το πει και να το επαναλάβει, δέχεται πλήρως την αρχή της απαλλαγής. Επαναλαμβάνω, αυτό το έχει επιβεβαιώσει η κυρία Άστον και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα, υπήρξαν διάφορες παρατηρήσεις για το ότι δεν τροποποιούμε το άρθρο 145 του δημοσιονομικού κανονισμού. Αλλά εδώ νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε για το ότι είναι η ίδια η συνθήκη στο άρθρο 319 παράγραφος Β που λέει ότι η απαλλαγή δίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολιτικά δίνεται απαλλαγή και σε άλλα όργανα. Και το ξέρουμε ότι αυτή είναι η πρακτική που ισχύει εδώ. Ναι λοιπόν πρόεδρε, τι είχα να σας πω. σχετικά με τα διάφορα στοιχεία που ανέπτυξαν οι συγκητές σας. Πιθανόν κάποια σημεία να μην ε, κάποια σημεία να μην τα έθιξα επαρκώς. Αν θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας πάντως. Ευχαριστώ. Κυρία Γκρέσλε. Σας ευχαριστώ. Εγώ δεν πιστεύω πλέον στον Άγιο Βασίλη, κύριε Γενική Διευθυντά. Είναι μάτιες όλες οι προσπάθειες εδώ και 8 χρόνια να με πείσετε περί της υπάρξεώς του. Η πρόταση που έχει τεθεί επιτάπητος από τη δική μας σκοπιά είναι ιδιαίτερα προβληματική. Δηλαδή, εάν η ευθύνη απόδοση λογαριασμών είναι μόνο θεωρητική, μπορούμε να πούμε εντάξει, λύσαμε όλα τα προβλήματα. Το πρόβλημά μας είναι ότι η απόκριση εκείνων που λαμβάνουν τις αποφάσεις από εκείνους οι οποίοι τις εκτελούν, αντιτίθεται στον ίδιο τον δημοσιονομικό κανονισμό. Η πρόταση Άστον φαίνεται σαν να μην έχουν λάβει καν υπόψη τα τελευταία 10-15 χρόνια των προσπαθειών της ε, Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Εμεί προσπαθήσαμε πάντοτε να εντοπίσουμε τις αδυναμίες της απόδοση λογαριασμών και έχουμε μπροστά μας τελικά ένα κείμενο όπου εντελώς ευθυνδιασμένοι αναγκαζόμαστε να τρίβουμε τα μάτια μας και να πούμε «Μα είναι δυνατόν, δεν έχετε καταλάβει απολύτως τίποτα». φαίνεται σαν να μην υπάρχει απολύτω καμία κατανόηση από μέρου σα για τα όσα έχει προσπαθήσει να εξηγήσει επί τόσα χρόνια η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού. Και έχω και ορισμένε ερωτήσει στην βάση του τι προσπαθούμε να επεξεργαστούμε. Δηλαδή και στην βάση τίνο εγγράφου, στη βάση προτάσεω Άστον ή στην βάση του συμβαστικού εγγράφου τη Ισπανική Προεδρία. Έγγραφο που σε κρίσιμα σημεία επιτείνει τις αδυναμίες του εγγράφου Άστον που ήδη είναι παραβίαση του ισχύοντος δημοσιονομικού κανονισμού και του ισχύοντος εργατικού δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που υπάρχουν λόγοι που είναι όπως είναι. Εφόσον πρόκειται να ιδρυθεί όργανο το οποίο θέλουμε να είναι νομικός ισχυρό, πώς ένα τέτοιο θεσμικό όργανο πώς θα διαμορφώσουμε θεσμικό όργανο το οποίο δεν προβλέπεται στις συνθήκες που δεν μπορεί να εμφανιστεί και στο δημοσιονομικό κανονισμό. Για παράδειγμα, το Συμβούλιο και ο πρόεδρος του Συμβουλίου είναι θεσμικά όργανα, δεν εμφανίζονται όμως στον δημοσιονομικό κανονισμό. Τίθεται λοιπόν θέμα της απαλλαγής. Ο κ. Σοντή θα μου πει ότι δεν υπάρχει νομική βάση γι' αυτό. Επομένως, ό,τι και να θεωρώ ότι ισχύει για την πολιτική απαλλαγή, πολιτικού χαρακτήρα απαλλαγή, πρέπει να υπάρχει και στο δημοσιονομικό κανονισμό. Πρέπει να καθίσουμε να επανορίσουμε δηλαδή τι σημαίνει δικαίωμα χορήγησης απαλλαγής και ποιες θα είναι οι συνέπειες εάν για παράδειγμα αρνηθούμε την απαλλαγή στην κυρία Άστον ή στον οποιοδήποτε διαδοχό της. Οι συνέπειες είναι απολύτως ασαφείς για την νομική φύση του εγγράφου που υποτίθεται ότι θα μας θέσει υπόψη η Ισπανική Προεδρία θα ήθελα να γνωρίζω κάτι. Δηλαδή περί τίνος πρόκειται. Επίσης διαβάζω το έγγραφο ότι μόνο η Κομισιόν μπορεί να υποβάλει προτάσεις. Και είχαμε διαφωνήσει με την Επιτροπή όταν μιλούσαμε για την Συμφωνία Πλαίσιο. Και τώρα στο έγγραφο της Ισπανικής Προεδρίας περιλαμβάνεται ότι η εκπρόσωπος έχει δικαίωμα πρωτοβουλίας και για την προγραμματισμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα προγραμματίζει αυτά και τα εκτελεί. Όμως στην πρόταση της Ισπανικής Προεδρίας το 8 αποκλείεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την διαμόρφωση ορισμένων προγραμμάτων όπως για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα. Δεν είχαμε επιρροή στον τρόπο που δαπανώνται 280 εκατομμύρια ευρώ στην πολιτική αυτή. Και τώρα το ποσό πολλαπλασιάζεται ως συνέπεια των προτάσεων αυτών να θέλετε να μας πουλήσετε τώρα αυτές τις προτάσεις ως βελτίωση είναι σαν να προσπαθείτε να μας πείσετε πράγματι για την ύπαρξη του Άγιου Βασίλειου. Να είσαστε σύντομοι οι επόμενοι, διότι έχουμε και άλλα θέματα στην ε, μυρισιά διάταξη. Ριβελίνη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να υποβάλω δύο ερωτήματα στον ε, Διευθυντή. Το πρώτο έχει ως εξής. Ίσως υπάρχουν ε, δυσκολίες στις μεταφράσεις. Αν ε, διαβάσουμε το άρθρο 50 στο αγγλικό, ιταλικό και γερμανικό κείμενο υπάρχουν ορισμένες αμφιβολίες. Ίσως θα πρέπει να ζητήσουμε μία πιο ε, σαφή μετάφραση για να μας ε, διασαφίσει το άρθρο 50 που είναι ζωτική σημασίας. Θα θέλαμε να ξέρουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσο δαπανάτε σήμερα για τις αντιπροσωπείες σας ανά τον κόσμο τι θα δαπανίσετε στο μέλλον. Αυτός ο αριθμός θα αφορά τις αντιπροσωπείες άμεσου ελέγχου ή και για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Αν δεν μας δώσει απαντήσεις η Επιτροπή, τότε γιατί γίνεται η όλη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, υπογραμμίσω τους ε, φόβους, να τονίσω τους ε, φόβους της κυρίας Γκρέσλε και θα ήθελα να διασαφηνίσουμε μιας διαπαντός αυτή τη διαδικασία απαλλαγής. Αυτό που μας οδηγεί σε συγχύσεις είναι ότι είχαμε πρακτικές απαλλαγές, απαλλαγής που δεν συμβαδίζουν με την ένωμη τάξη. Γι' αυτό είχα ζητήσει μία ε, νομοθετική μελέτη. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβουμε υπόψη ότι είναι νομικό πρόσωπο. Γι' αυτό εμείς θα πρέπει να χορηγούμε απαλλαγή, μία απαλλαγή ανανομικό πρόσωπο. Σήμερα λέμε δίνουμε απαλλαγή, χορήγουμε απαλλαγή στο τάδε θεσμικό όργανο, στην Επιτροπή Περιφερειών και ούτω καθεξής. Αυτή η εξωτερική υπηρεσία είναι μια υπηρεσία και σύμφωνα με αυτά που αναφέρει η συνθήκη και ως εκτελεστικό της Ένωσης η Επιτροπή χορηγεί, υποβοηθά μάλλον στην απαλλαγή εκτελεστικό δηλαδή όργανο είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά είναι υπεύθυνη για το σύνολο του προπολογισμού. Ακούγοντας τους μεν και τους δε, νομίζω ότι θα πρέπει να υποβάλουμε ε, τροπολογίες. Ε, εμείς έχουμε την, ε, το δικαίωμα ελέγχου επί, επί όλων των οργάνων και θα πρέπει το θέμα να διευκρινιστεί και σε έναν κανονισμό. Πρόκειται όμως για μια υπηρεσία σου αλλά είναι, δεν είναι παρά μόνο μία υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι νομικό πρόσωπο. Κάλφιν. Ευχαριστώ. Δύο σύντομες ερωτήσεις. Προς τον κύριο Ζων Κύριε Γενική εάν ένα ευρωβουλευτή θέλει να θέσει το ερώτημα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των ταμείων των χρημάτων που δαπανώνται για παράδειγμα στην Γάζα ή στο Αφγανιστάν, ποιον πρέπει να ερωτήσει. Δεύτερο, θεωρείται ότι η μετακίνηση ορισμένων στελεχών του προσωπικού από την Κομισιόν και το Συμβούλιο προ την ε, Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων θα συμβαδίσει με τον προπολογισμό των διοικητικών αυτών δαπανών και δεν μιλώ βέβαια για το, προσωπικό, το πρόσθετο προσωπικό το οποίο θα προέρχεται από τις χώρες μέλη. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο δίνω στον Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Yeah. Ευχαριστώ. Σε σχέση με το ερώτημα του κυρίου Ριβελίνη για το άρθρο 50 του Δημοσιονομικού Κανονισμού εδώ είναι μια δυνατότητα που παραμένει ανοιχτή. Έτσι το επιθυμούσαμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να διαχειριστεί η ίδια ορισμένα ε, διοικητικά κονδύλια παρά να τα αναθέσει κατά εξουσιοδότηση. Δηλαδή η Επιτροπή σε εισαγωγικά ε, διαθέτει τα κονδύλια στα άλλα θεσμικά όργανα για διοικητικές δαπάνες. Υπάρχει ένα ειδικό σχήμα για την διαχείριση ορισμένων υπηρεσιών. Αν θέλουμε να ενοποιήσουμε τη διαχείριση και να την κάνουμε πιο αποτελεσματική, θα πρέπει να έχουμε μια κατάσταση όπου η Επιτροπή δεν μεταφέρει όλα τα κονδύλια στην, ε, εξωτερική, στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης, αλλά μπορεί να δράσει μαζί με αυτή την υπηρεσία. Αυτό το σενάριο δεν ισχύει αλλά είναι μία δυνατότητα που διαγράφεται. Όσον αφορά τις πράξεις ε, εξουσιοδότηση, θα ήθελα να είμαι απόλυτα σαφής. Υπάρχει ένας προϋπολογισμός για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης με έναν ε, προπολογισμό για το σύνολο των αντιπροσωπιών. Εκεί υπάρχει προσωπικό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα συμμετάσχει στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης, δηλαδή όλο το προσωπικό εκτός από τους επικεφαλείς αντιπροσωπιών και το πολιτικό, το προσωπικό. Το υπόλοιπο επίσης προσωπικό που θα ασχοληθεί με την εμπορική διαχείριση, γενομικό έλεγχο, συνεργασία σε επιστημονικά θέματα και οι υπάλληλοι της Κομισιόν που διαχειρίζονται συνεργασία και την ανάπτυξη. Αυτό το προσωπικό είναι προσωπικό της Κομισιόν, το οποίο ε, υπόκειται στην Κομισιόν, βρίσκεται στον, ε, και υπόκειται στον ε, διοικητικό Προϋπολογισμό της Επιτροπής. Άρα δεν θα επέλθει καμία αλλαγή, διότι η Επιτροπή ε, εφορμάζοντας αυτή την, πολιτική, την αναπτυξιακή της πολιτική, θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σε σχέση με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Η απάντηση θα σας δοθεί όταν η κυρία Άστον, η Κομισιόν και η κυρία Άστον θα υποβάλουν τον διορθωτικό προϋπολογισμό. Στο Συμβούλιο πολλές αντιπροσωπείες θέλουν να τηρηθεί η αρχή της ε, δημοσιονομικής ουδετερότητας. Όσον αφορά το ερώτημα του κυρίου Κάλφιν για την διαχείριση των κονδυλίων στη Γάζα, εάν τα κονδύλια αυτά την χάνουν μιας διαχείρισης μέσω ε, ε, επιχειρησιακών δαπανών, τότε η Επίτροπος ή ο Επίτροπος υπεύθυνο για θέματα συνεργασίας είναι υπεύθυνο για την ε, καλή διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Και αυτό γίνεται σε συνεργασία με την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής αλλά ο αρμόδιος επίτροπος είναι υπεύθυνος, ο επίτροπος ο οποίος ασχολείται με την αναπτυξιακή βοήθεια, με θέματα ανάπτυξης. Και βεβαίως πίσω από όλα αυτά είναι το Διευθυντήριο των Επιτρόπων. Όσον αφορά τώρα το προσωπικό, νομίζω ότι απάντησα στο ερώτημα ήδη, ε, απαντώντας στον κύριο Ριβελίνη, δηλαδή Όσον αφορά τους υπαλλήλους οι οποίοι υπάγονται στην Κομισιόν, θα εξακολουθήσουν να υπάγονται στην Κομισιόν και η δημοσιονομική κατάσταση δεν θα αλλάξει επειδή δημιουργείται αυτή η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Όσο αφορά την κυρία Άστον, σε συνεργασία με την Κομισιόν θα υποβάλει προτάσεις με στα πλαίσια του διορθωτικού προπολογισμού που θα ε, υποβάλει η Επιτροπή εν ευθέτω χρόνο. Λαμβάνω υπόψη τις ε, σκέψεις σας σε σχέση με θέματα απαλλαγής. Σε αυτό το στάδιο δεν θα ήθελα να κάνω σχόλια, ιδιαίτερα σχόλια, σε σχέση με αυτά που ανέφερε. Πολύ ενδιαφέρουσα, εν πάση η ερώτησή του. Σα ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο σημείο 8 της σημερινή διάταξη, δηλαδή τροποποίηση του κανονισμού 1605 2002 του Συμβουλίου σε σχέση με τον δημοσιονομικό κανονισμό ε, που εφαρμόζεται στο Γενικό Προπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο κύριος Ριβελίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος ε, για τη δεύτερη αυτή παρένθεση στην Επιτροπή Κοντ σε σχέση με τον κανονισμό του Συμβουλίου για τον δημοσιονομικό κανονισμό που αφορά το γενικό προϋπολογισμό. Αλλάζουμε λοιπόν το δημοσιονομικό κανονισμό μετά από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Άρα στα, στα πλαίσια του τριετούς ελέγχου δημιουργείται μια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης οι περισσότερες τροποποιήσεις της πρότασης έχουν σαν στόχο την δημοσιονομική διαδικασία όπως ορίζει η συνθήκη. Και για αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την απόψη 17 Μαρτίου 2006 της Διαθεσμικής Συμφωνίας για την Δημοσιονομική Πειθαρχία. Και γι' αυτό αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να εισαχθούν στο κείμενο του δημοσιονομικού κανονισμού. Ως προς την αρμοδιότητα της ΚΟΝΤ προβλήθηκε μία πρόταση τροποποίησης για να αλλάξουμε το 146.2 για τις τροποποίησεις που απορρέουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Σύμφωνα με το άρθρο 318 η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μία έκθεση αξιολόγησης των δημοσιονομικών της Ένωσης με βάση τα αποτελέσματα. Η πρόταση τροποποίησης μιλά για αξιολόγηση μαζί με τα έγγραφα τα οποία θα επισυναυθούν από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Υπάρχουν όμως και άλλες πτυχές που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Πρώτον, πέρα από τα ερωτηματικά που προανέφερα σε σχέση με την τροποποίηση του άρθρου 49 του Δημοσιονομικού Κανονισμού για τη, τα κονδύλια που εντάσσονται στον προϋπολογισμό και για τις ειδικέ δράσεις και ιδιαίτερα για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, εδώ επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να αποφανθεί η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα να σας επισύρω την προσοχή στο γεγονός ότι η Κομισιόν δεν μας έκανε υποδείξεις για τις μελλοντικές διατάξεις σε θέματα ελέγχου και λογιστικών αλλαγών για την επικαιροποίηση του προϋπολογισμού, όπως ορίζει το άρθρο 317. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρκέστηκε να αναφέρει στην αιτιολογική έκθεση ότι οι διατάξεις αυτές μαζί με το, το 44 που αφορά την δημοσιονομική διαχείριση θα αποτελέσουν αντικείμενο εμβαθυμένης ανάλυσης με βάση την τριετή αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού. Αυτές οι διατάξεις είναι ύψης της σημασίας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει σαφής λογοδοσία των κρατών μελών ως προς την διαχείριση των κονδυλίων. Άρα η πρότασή μου, όπως είπα και για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η πρότασή μου είναι απόλυτα σαφής, διότι θα πρέπει να γίνεται ευφυής χρήση των δημοσίων πόρων, να υπάρχει ποιότητα στις ε, νομοθετικές μας πράξεις. Και γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το δημοσιονομικό κανονισμό μαζί με την πρόταση τροποποίησης, τη γενικότερη ε, πρόταση τροποποίησης του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να προσαρμοστούμε στα δεδομένα της συνθήκης της Λισαβόνας, στα πλαίσια της τριετούς αναθεώρησης. Βεβαίως, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια πιο ομοιογενή ε, νομοθετική πρόταση, η οποία να διασαφινιστεί περισσότερα. Το λόγο έχει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Παρακαλώ. Euh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα τον εισηγητή, τον κύριο Ριβελίνη, και θα ήθελα γι' αυτό να πω δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, σε σχέση με μια ταυτόχρονη αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και τριετή και βάσει τις συνθήκες της Λισαβόνας. Πρόεδρε, επήγει το θέμα. Πρέπει να πάρουμε γρήγορα απόφαση όσον αφορά την δημιουργία και λειτουργία της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Είμαστε σε ένα στάδιο όπου ο κόσμος ολόκληρος έχει στραμμένα τα μάτια του απάνω μας. Προσπαθεί να δει τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό λοιπόν η υπηρεσία αυτή να μπορέσει να αρχίσει να λειτουργεί πλήρως όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και γι' αυτό ακριβώς εξάλλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμφωνία με την ύπατο εκπρόσωπο υπέβαλε μια ξεχωριστή πρόταση. Όσο ο δημοσιονομικός κανονισμός και ο προπολογισμό και αποφάσεις για το προσωπικό δεν έχουν ληφθεί, η υπηρεσία αυτή δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Είναι όμως χρέος όλων μας. Να φροντίσουμε να πάνε τα πράγματα γρήγορα. Φυσικά και πρέπει να γίνει η πολιτική συζήτηση και γίνεται. Αλλά πρέπει συγχρόνως να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα. Όσον αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας, οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι γνωστές. Εμείς θέλουμε τεχνικής φύσεως προσαρμογή των ε, διατάξεων που υπάρχουν στην διοργανική συμφωνία. Μόνο των τεχνικών διατάξεων γνωρίζοντας ότι προτιμήσαμε για άλλες πιο περιορισμένες όμως διατάξεις, πολύ λίγες που είναι την συνθήκη να περιμένουμε την αναθεώρηση την τριετή που θα καλύπτει ένα ευρύτερο πεδίο. Η πρόταση αυτή της Επιτροπής, όπως ξέρετε Πρόεδρε, θα εγκριθεί εφόσον όλα πάνε καλά από το Σώμα των Επιτρόπων στις 26 Μαΐου που μας έρχεται. Πιστεύω λοιπόν ότι ό,τι λείπει μέχρι τώρα, όπως λέει και ο κύριος Ριβελίνη, το θέμα της δήλωση για παράδειγμα, είναι πράγματα τα οποία θα υπάρχουν. Και έτσι θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Γκρέσλε. Λίγες φράσει Μόνο αν και σημειώνω ότι ο γενικό διευθυντή τίνει να μην απαντά τι ερωτήσει μου. Μέχρι τώρα οι κινήσεις αυτές έχουν γίνει σε βάρος μας. Οι προτάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα για την, για την ε, Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων είναι σε βάρος του Κοινοβουλίου. Το πρόβλημα είναι ότι όσο δεν γνωρίζουμε και μιλούμε για μεταφορές, όσο δεν γνωρίζουμε ποια μορφή θα λάβει η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, πρέπει να προσέξουμε ώστε στην πρώτη ανάγνωση να μην κάνουμε πράγματα τα οποία θα μετανιώσουμε στη δεύτερη ανάγνωση. Γι' αυτό όλες αυτές οι προτάσεις αναθεωρήσεων αναφέρονται στα ίδια άρθρα. Γι' αυτό είναι σκόπιμο να αναμείνουμε να δούμε τι θα τεθεί επιτάπητος. Κύριε Γενικέ Διευθυντά, θα ήταν ωραία να μας είχατε απαντήσει για τις εθνικές δηλώσεις. Από την πρώτη ίδια αναθεώρηση να είχατε υποβάλει κάτι. Στην πρώτη αναθεώρηση βγαίνει η Επιτροπή και ζητάει κάτι από εμάς. Στην δεύτερη το Συμβούλιο και στην τρίτη το Κοινοβούλιο από το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Αλλά με ποια δυνατότητα πίεσης. Ο κ. Ριβελίνη έχει δίκιο. Ας περιμένουμε και ας τα προωθήσουμε τα πράγματα αυτά εν τέλει με τη δική μας ταχύτητα και με τρόπο προσεκτικό. Περνάμε στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης η αντιπροσωπεία στην Ελλάδα από αύριο μέχρι τις 29 Απριλίου. Θα πρέπει να γίνει μία ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη της Επιτροπής για να δούμε ποια είναι τα σημεία τα οποία είναι τα πλέον κρίσιμα που θα αντιμετωπίσει τις επόμενες μέρες η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού στην Ελλάδα. Έχετε το υλικό ενώπιόν σας. Τέσσερα είναι τα κρίσιμα σημεία. Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, συστήματα διαχείρισης των διαφορετικών ταμείων, το Ταμείο Ελληνικής για την Ελλάδα, η ανεξαρτησία της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας και η παρουσία της Όλαφ στην ε, Ελλάδα. Θα γίνει μια συζήτηση με την Επιτροπή μέχρι τις 18 και 10 και το τελευταίο ημίωρο με τα μέλη της ΟΛΑΦ και κλεισμένων των θυρών. Ποιος θα ήθελε να παρέμβει, έχετε το λόγο. Κάρλο Πετινέλη, DG Employment. Κάρλο Πετινέλη. Θέλω να αναφερθώ στο πρώτο ε, κατάλογο. Να σας πω ότι εμεί ε, δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα για την Ελλάδα. Όλοι οι έλεγχοι που έχουμε κάνει έδειξαν ότι υπάρχει ένα περιθώριο σφάλματος αρκετά χαμηλό και δεν υπάρχουν ε, σοβαρά συστημικά προβλήματα. Οι ελληνικές αρχές κάθε φορά που βρίσκανε προβλήματα κάνανε οι ίδιες τις διορθώσεις και όσον αφορά το λειτουργικό πρόγραμμα έχει μπει υπό τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Για την περίοδο 2000-2006 κάναμε 10 ελέγχους ε, στα 20 προγράμματα. Και τα προβλήματα ήταν πολύ μικρά, με διορθώσεις που είχαν κάνει οι ίδιες ελληνικές αρχές της τάξης των 14 εκατομμυρίων. Ξέρουμε ότι το ελεγκτικό συνέδριο στα πλαίσια της ΔΑΣ 2007 και 2008 πήγε στην Ελλάδα για τα λειτουργικά προγράμματα αλλά δεν ε, κατέληξαν σε σφάλματα όσον αφορά τη δήλωση εξοπιστίας ΔΑΣ και ούτε έγιναν σημαντικές ε, επικρίσεις για τα συστήματα ελέγχου. Το ίδιο και την περίοδο προγραμματισμού του Κοινωνικού Ταμείου 2007-2013. Και εδώ τα προγράμματα ξεκίνησαν. Η Ελλάδα δεν ήταν από τις χώρες που είχαν καθυστερήσει για το Converse Assessment, για την εφαρμογή δηλαδή των συστημάτων ελέγχου, είχαν όλα γίνει μέχρι τα τέλη του 2009. Άρα τα πράγματα προχωράνε κανονικά. Μπορούμε συνεπώς να έχουμε θετικό συμπέρασμα. Όσον αφορά την απλοποίηση, οι ελληνικές αρχές αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα της δήλωσης του έμεσου ε, εξόδου κατά αποκοπή. Ζητήσαμε λοιπόν συμπληρωματικές επεξηγήσεις και περιμένουμε ακόμα τις απαντήσεις από τις ελληνικές αρχές. Εδώ δίπλα μου έχω τον συνάδελφο του Περιφερειακού Ταμείου. Ευχαριστώ. Θέλω να προσθέσω και εγώ κάποια στοιχεία για να τα ακούσουν οι ευρωβουλευτές. Πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης και ελέγχου το οποίο είναι σχετικά περίπλοκο. Ξέρετε ότι τα προγράμματα τίθενται σε εφαρμογή σε πέντε περιφέρειες και υπάρχουν 14 προγράμματα, πέντε περιφερειακά και 8 τομεακά. Το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου έχει μία ενιαία αρχή για άδεια, μία ενιαία αρχή για τον έλεγχο και ένα όργανο συντονιστικό για το συντονισμό. Ενία πάλι. Οι περιφέρειες είναι οι ενδιάμεση. Θέλω εδώ να υπογραμμίσω τρία στοιχεία. Πρώτον, ότι είναι περίπλοκο το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Οι ελληνικές αρχές μελετούν συστήματα απλοποίησης, ιδιαίτερα για να υπάρξει καλύτερος συντονισμός και πιο αποτελεσματική διαχείριση. Θέλω εδώ να επενθυμίσω ότι η εφαρμογή των προγραμμάτων για την νέα περίοδο 2007-2013 στην Ελλάδα πάει αργά. 4% μόνο έχει απορροφηθεί μέχρι τώρα Το κονδυλίων, ένα δισεκατομμύριο δηλαδή. Και αυτό οφείλεται κυρίως σε δυσκολίες που υπάρχουν όσον αφορά τα δημοσιονομικά της χώρας, αλλά και επειδή οι διαδικασίες είναι περίπλοκες. Επίσης δεν υπάρχουν και όριμα προγράμματα τα οποία να είναι έτοιμα να τεθούν σε εφαρμογή. Ένα δεύτερο στοιχείο που πιστεύω ότι είναι σημαντικό εδώ είναι ότι υπάρχουν διάφορα προβλήματα όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις. Τις προηγούμενες χρονιές διαπιστώσαμε αδυναμίες στη διαχείριση και στον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων. Οι ελληνικές αρχές ε, ετοιμάζουν προγράμματα ενημέρωση ελέγχου, πολύ πιο περίπλοκα για αυτό το θέμα. Για την προηγούμενη περίοδο πάντως η Ελλάδα χρειάστηκε να περάσει από, διορθώσει από οικονομικές σε ένα μεγάλο βαθμό. 580 εκατομμύρια για το ΦΕΝΤΕΡ και 23 εκατομμύρια για το Ταμείο Συνοχής. Και όλα αυτά εξαιτία διαφόρων ατασταλιών που παρατηρήθηκαν κυρίως όσον αφορά τον οικοδομικό τομέα, τα έργα, έργα υποδομών. Ο κίνδυνος για τις δημόσιες αγορές σήμερα είναι περιορισμένος. Αλλά, όπως έλεγα, εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις. Ένα τελευταίο σημείο που θέλω εδώ να υπογραμμίσω έχει να κάνει με το Ταμείο Αλληλεγγύης. Η Ελλάδα ζήτησε χρηματοδότηση 6 φορές από το 2002. Από τότε που άρχισε δηλαδή να ισχύει το Ταμείο Αλληλεγγύης 2, έγιναν αποδεκτές. Κυρίως μετά τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές. Δύο συζητιώνται τώρα, δεν έχουμε αποφασίσει και άλλες δύο απορρίφθηκαν. Δύο λοιπόν ε, φορές χρησιμοποιήθηκε το Ταμείο Αλληλεγγύης για την Ελλάδα. Όσον αφορά την καθυστέρηση της εφαρμογής, αυτό είναι το τελευταίο μου, οφείλεται στο ότι οι ελληνικές αρχές δεν χρησιμοποίησαν όλες τις δυνατότητες που είχαν. Υπάρχει ένα ταμείο επενδύσεων που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και το οποίο δεν χρησιμοποιήθηκε. Το Ταμείο αυτό προσφέρει δυνατότητες και ευκαιρίες πολύ μεγάλες. Κυρίως για επενδύσεις στις μικρές και μεσές επιχειρήσεις, αλλά και για μεγαλύτερα έργα. Στα, στο θέμα των απορριμμάτων των πόλεων. Να λοιπόν, μια σύντομη παρουσίαση των κυρίων σημείων που θα μας απασχολήσουν στην επίσκεψη στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλοι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα ήθελα να λάβουν το λόγο. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Πρόστε έναν. Είμαι η αναπληρωτής διευθυντής στην Γενική Διεύθυνση Άγκρη. Ε, θα ήθελα να σας μιλήσω για το σύστημα Άγιαξ που ισχύει στην Ελλάδα. Όπως ξέρετε υπάρχει το σύστημα Άγιαξ το οποίο ισχύει από το 98 σε κάθε κράτος μέλος και είδαμε μετά από 10 χρόνια ότι το σύστημα είναι ελληματικό στην Ελλάδα. Το, το 2010 ορίσαμε ένα πρόγραμμα δράσης ε, για την Ελλάδα έτσι ώστε να διορθωθεί η κατάσταση από το 2008. Και στις αρχές του 2009, μετά το 2008, είδαμε ότι για τέσσερα βασικά σημεία του προγράμματος ε, δράσης η Ελλάδα ανταποκρίθηκε. Το LPAS όμως, το Partial Identification System, είναι ένα σύστημα με το οποίο μπορούμε να ορίσουμε τα αγροτεμάχια. Η Ελλάδα μας έδωσε νέες φωτογραφίες, ψηφιακές φωτογραφίες χαρτογράφησης όπου έχουμε ε, τα αγροτεμάχια που υπάγονται και αυτά που δεν υπάγονται. Αυτό από το Φεβρουάριο του 2009. Επίσης διαπιστώσαμε ότι το LPS ισχύει και μπορεί να ισχύσει, υπάρχει το λογισμικό και όλες οι υπηρεσίες ε, καταβάλουν κάθε προσπάθεια, ακόμα και τα συνδικάτα, οι πάντες έχουν ε, προσβασιμότητα, έχουν πρόσβαση σε αυτό το νέο σχέδιο, το οποίο έχει στε από επιτυχία. Τότε η κυρία Φίσε Μπόλ σας είχε αποστείλει στοιχεία με τα αποτελέσματα. Η Επίτροπος και αποστήλαμε φωτογραφίες. Έχετε φωτογραφίες, δύο σειρές φωτογραφιών, δύο φορές από τρεις στο παράρτημα. Έχετε το παλαιό LPAS και το νέο LPAS, δηλαδή το σύστημα κατάτμισης αγροτεμαχίων. Και βλέπετε τα αγροτεμάχια που έχουν οριστεί με κίτρινο χρώμα, είναι τα μη επιλέξιμα. Αυτό είναι το σημείο κίνησης του ΕΛΠΕΙΕΣ που ισχύει από το 2009. Κατά το πρώτο έτος εφαρμογής κάθε αγρότης θα πρέπει στα πλαίσια αυτών των μπλοκ να ορίσει το δικό του αγροτεμάχιο και αυτή η εργασία βρίσκεται στο πρώτο έτος εφαρμογής. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει η πρώτη χαρτογράφηση το Μάιο του 2009 και μετά βλέπουμε μόνο τις τροποποίησεις. Αλλά η μεγάλη, ε, το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας έχει επιτελεστεί και είδαμε ότι οι αγρότες δεν ήρθαν εγκαίρως και μπορούμε να αναρωτηθούμε γιατί. Ε, φοβούνται αυτό το σύστημα ε, βρισκόμαστε στην προεκλογική, σε προεκλογική περίοδο το μήνυμα δεν ήταν σαφές. Ε, δηλαδή ότι όποιος αγρότης δεν προβεί σε δήλωση δεν μπορεί να τύχει και επιδότησης, δηλαδή δεν έχει δικαίωμα επιδότησης. Εν πάση περιπτώσει το φθινόπωρο διαπιστώσαμε ότι τα αιτήματα επιδότησης δεν εισήχθησαν καιρος και τότε παρενέβη η Κομισιόν και ορίσαμε μια νέα ημερομηνία ε, λέγοντας τους αγρότες ότι αν δεν υποβάλουν ε, το αίτημά τους εγκαίρως δεν θα μπορέσουν φέτος να τύχουν επιδότησης. Μετά από αυτό ορίστηκε η ημερομηνία στα τέλη Ιανουαρίου του 2010 και είδαμε ότι ε, πράγματι με τη νέα κυβέρνηση είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή αυτό τι σημαίνει. Ότι το 2009 ότι το LPS λειτουργήσε αλλά με σημαντικές καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις οι οποίες δεν σχετίζονται με το νέο σύστημα αλλά ε, από το ότι δεν ε, υπήρξε μία σωστή κατευθυντήρια γραμμή. Τώρα που ορίσαμε το 2009, το οριοθετήσαμε σωστά, είμαστε σίγουροι για το 2010. Υπέβαλα δύο ερωτήματα στους Έλληνες συναδέλφους. Καταρχήν να μου κάνουν μία πρόβλεψη των αγροτεμαχίων όπου για τα οποία θα πρέπει να προσέλθουν ε, οι αγρότες, γιατί μερικοί δεν προσήλθαν εγκαίρως, δηλαδή προσήλθαν μεν, αλλά δεν αναγνώρισαν σωστά τα αγροτεμάχια τους. Και βεβαίως κάθε χρόνο επέρχονται και αλλαγές. Έγινε αυτή η εκτίμηση και μέχρι τις 15 ε, Μαΐου ε, είναι η προθεσμία, δηλαδή Μάρτιος με 15 Μαΐου, μπορεί να γίνει θεωρητικά. Η Ελλάδα όμως είναι οργανωμένη για να κάνει κάτι τέτοιο, να μην αντιμετωπίσει τα, τα προβλήματα του προηγούμενου έτους. Οι Έλληνες εφήβραν ένα σύστημα όπου, όπου συνεργάζονται όχι πια με τα συνδεκάτα, αλλά με τις τράπεζες και τα πανεπιστήμια, δηλαδή θέλαν να εφεύρουν εκ νέου ένα σύστημα, ένα νέο σύστημα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς τους είπαμε να συνεργαστούν με τα συνδικάτα, τα καλύτερα συνδικάτα και τις υπηρεσίες ανάπτυξης. Δηλαδή κάτι τέτοιο είναι δυνατό να επιτευχθεί και η Ελλάδα αποφάσισε ότι για τα μικροετήματα, τα μικροετήματα δεν γίνονται ε, αποδεκτά, άρα γίνεται μία διάκριση μεταξύ του πραγματικού όγκου εργασίας και των επιμέρους ζητημάτων ίσονος σημασίας, τα οποία δεν πρέπει να μας απασχολήσουν. Η Συνάδελφοι, επιτόπου τον Ιούνιο θα δούνε κατά πόσο λειτουργήσε το σύστημα και είναι ποιοτικό καλό, αλλά το LPS, το πρόγραμμα δράσης, ε, τηρήθηκε, ήταν πολύ καλό. Στο πρώτο έτος εφαρμογής γνωρίσαμε μια μεγάλη καθυστέρηση που θα έχει επιπτώσει στην εκαθάριση λογαριασμών. Ε, διορθώσαμε εγκαίρως τα σφάλματα και τώρα ζητάμε από τις ελληνικές αρχές να εξασφαλίσουν την καλή διαχείριση για το 2010. Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Ματισόφ. Είμαι επικεφαλής στη Eurostat της Νομικής Υπηρεσίας και προτείνω σύντομα να σας παρουσιάσω αυτό που έχουμε ετοιμάσει για το ελληνικό στατιστικό σύστημα από πλευρά δηλαδή ανεξαρτησίας και ακαιρεότητα. Ξέρετε πολύ καλά, μετά τα πρόσφατα γεγονότα από τον Οκτώβριο, όταν έγινε αναθεώρηση των στατιστικών δεδομένων όσον αφορά τις ε, μεγάλες αναθεωρήσεις, το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ετοιμάσει έκθεση για τα προβλήματα που τίθενται όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία από την Ελλάδα που ενέκρινε η Επιτροπή τον Ιανουάριο που μας πέρασε. Στην έκθεσή της αυτή η Επιτροπή παρουσιάζει νομίζω εκτενώς τα προβλήματα μεθοδολογίας που βρήκαμε στην Ελλάδα και που έχουν να κάνουν με δύο προβλήματα. Το ένα είναι μεθοδολογικές δυναμίες και τεχνικές διαδικασίες που δεν είναι ικανοποιητικέ και από την άλλη παραλήψεις πιο σοβαρές του ίδιου του συστήματος, του συστήματος μέσα από μια διαχείριση που δεν είναι ικανοποιητική, ούτε οι διαδικασίες είναι αρκετά σαφείς, ούτε ο τρόπος χειρισμού που γίνεται. Το Συμβούλιο Κοφίν λοιπόν του Ιανουαρίου ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσει τις προσπάθειές της για συνεργασία με τις ελληνικές αρχές. Προκειμένου να ενισχυθεί το ελληνικό στατιστικό σύστημα. Ζήτησε λοιπόν και από την Επιτροπή και από τις ελληνικές αρχές να υποβάλουν ένα σχέδιο δράσης. Το σχέδιο αυτό δράσης εκπονείται επί του παρόντος. Θα πάει στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή την επόμενη εβδομάδα και στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ 18 και 19 Μαΐου. Στο μεταξύ η Ελλάδα έκανε πολλές προσπάθειες ενέκρινε ένα νέο στατιστικό νόμο που δημιουργεί μια νέα στατιστική αρχή στην Ελλάδα που είναι ανεξάρτητη αρχή και που χέρι μια πλήρους επαγγελματικής ανεξαρτησίας από τις 9 Φεβρουαρίου κανονικά αλλά πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή. Υπάρχει και η διαδικασία επιπαραβάση της Επιτροπής βάρος της Ελλάδας μετά από την μεγάλη αναθεώρηση των ε, αριθμητικών στοιχείων του Οκτωβρίου, των στατιστικών δεδομένων και την Παρασκευή που μας πέρασε πήραμε την απάντηση από τις ελληνικές αρχές στο, στην επιστολή προειδοποίησης που στείλαμε και αναλύουμε την απάντηση αυτή. Κάτι άλλο που θέλω να σας πω είναι η πρωτοβουλία που πήρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να ενισχύσει τις αρχές της Eurostat στον έλεγχο και στην επαλήθευση της ποιότητας των δεδομένων, των στατιστικών δεδομένων που μας στέλνουν τα κράτη-μέλη. Και υπάρχει το ανακοινωθέν τύπου της Eurostat για τις κοινοποίησεις ε, στην Ελλάδα. Της πέμπτης που μας πέρασε, όπου η Eurostat μιλάει πάλι για την ποιότητα των στατιστικών δεδομένων που έχει διαθέσει η Ελλάδα. Όλα αυτά για να σας πω ότι η συνεργασία με τις ελληνικές αρχές ε, πηγαίνει προς την κατεύθυνση ενίσχυσης του στατιστικού μηχανισμού. Και σίγουρα η επίσκεψη της αντιπροσωπείας σας στην Ελλάδα θα επαληθεύσει τις διαθέσεις αυτές των ελληνικών αρχών να βελτιώσουν τον στατιστικό μηχανισμό. Η κυρία Γκρέσ. Ακούγοντας όλα αυτά τα ωραία, μου φαίνεται ότι δεν είναι και απαραίτητο καν να πάμε. Όλα είναι εντάξει. Ε, εγώ νομίζω ότι πρόκειται για ένα μέγα ε, πρόβλημα, όπως ένα μέγα πυρηνικό ατύχημα θα έλεγα, στη, αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς είναι δυνατόν να έχει διαρκέσει 13 χρόνια μέχρι να φτάσουμε με το IAX να έχουμε ένα αποτέλεσμα που να μπορούμε να δείξουμε. Κάνετε εσείς κάποια επιφύλαξη και αν όχι γιατί. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να έχει ένα περιθώριο σφάλματος 3% που το βρίσκω εκπληκτικά χαμηλό, που δείχνει ότι υπάρχουν και σφάλματα στο ίδιο το σύστημα. Το θέμα που τίθεται είναι τι θα πρέπει να κάνουμε. Ασφαλώς και σας είμαστε και προσωπικά ευγνώμονες, γιατί χωρίς την προσπάθειά σας δεν θα είχαν υπάρξει οι πρόοδοι αυτές και χωρίς την προσπάθεια της κυρίας Φίσερ φαίνεται καθαρά ότι όταν αναλαμβάνει αποφασιστικά δράση η Κομισιόν, αυτό αποφέρει αποτελέσματα. Και η Ευρωστάτ έκανε πολλά πράγματα. Προς τον εκπρόσωπο της Ευρωστάτ έχω την ερώτηση γιατί οι επιφυλάξεις σας δεν ελήφθησαν υπόψη. Εγώ δεν τις γνώριζα τις επιφυλάξεις αυτές. Και εάν είχαν γίνει γνωστέ οι επιφυλάξει αυτέ για τα ελληνικά στατιστικά στοιχεία, ποιο θα έπρεπε τότε να αναλάβει δράση. Και επίση, εάν υπάρχουν επιφυλάξει σχετικά με τον προπολογισμό του 2009. Ο κ. Ζοντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρεμβαίνω για το τελευταίο αυτό θέμα, δηλαδή την ποιότητα των στατιστικών στοιχείων. Κάπου με ενοχλεί ο όρος στατιστική. Για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερα να μιλάμε για προβλήματα χορήγησης δημοσιονομικών πληροφοριών. Υπάρχουν οι οργανισμοί στατιστικής, η Ευρωστάτ που παρεμβαίνει. Μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένα πρόβλημα της δημόσιας ενημέρωσης για στατιστικά θέματα. Ο κόσμος, οι πολίτες έχουν όλο και περισσότερο την εντύπωση ότι γίνεται κακοδιαχείριση. Δεν μιλώ τώρα για σύγκριση με την ιδιωτική σφαίρα. Δίνουμε τώρα ιδιαίτερο βάρος στην περίπτωση της Ελλάδας διότι υπάρχουν τα μεγάλα ελλείμματα. Αλλά η ποιότητα των δημοσιονομικών πληροφοριών όλων των χωρών μελών και της δικής μου θα μας εξέπλητε. Εγώ πάντως εκπλήσωμαι για το γεγονό ότι στο έγγραφο δεν γίνεται παρέμβαση των εθνικών ελεγκτικών συνεδρίων, δεν περιλαμβάνεται τέτοια, που θα ήταν χρήσιμο τα έγγραφα σχετικά με δημοσιονομικές πληροφορίες, με όλων των ειδών της στατιστικές κτλ, να συμπεριλαμβάνεται σε αυτά και μια βεβαίωση για την αξιοπιστία των λογαριασμών αυτών. Ακόμα και τώρα που θα είναι υποτίθεται ανεξάρτητη η αυτή αρχή στην Ελλάδα. Το ίδιο και οι εθνικοί βουλευτές, οι οποίοι οφείλουν να ελέγχουν την εκτελεστική εξουσία στις χώρες μέλη. Υπάρχει εδώ, ανοίγεται εδώ ένα πεδίο συνεργασίας Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων για να εξασφαλιστεί μια καλύτερη ποιότητα των πληροφοριών αυτών, την οποία έχουμε ανάγκη για την ε, χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών έργων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούγοντας την ε, παρουσίαση και κοιτώντας και τα κείμενα που έχουν ετοιμαστεί για την αυριανή αναχώρηση, έχω την αίσθηση ότι η Επιτροπή, με κάπως πομπόδι τρόπο, ξεχνάει την κρίση που περνάει η Ελλάδα σήμερα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, βγάζοντας συμπεράσματα από το ελληνικό παράδειγμα, πιστεύετε ότι έχετε τη δυνατότητα να προειδοποιήσετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για κινδύνους που ενδεχομένως υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες από την Ελλάδα. Δεν παίρνουμε κάποιο μάθημα, δεν μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα ή για άλλη μια φορά με τρόπο έτσι πομπόδι θα μιλήσουμε κάποτε αργότερα στο μέλλον για μια άλλη χώρα που θα περάσει από τέτοια προβλήματα. Μακάρι όχι. Αλλά αν υπάρχει μια Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού, αυτό το ρόλο πρέπει να παίζει. Πώς μπορούμε να προλάβουμε τέτοιους κινδύνους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Σκέλη. Ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις για τους αξιότιμους συναδέλφους της Κομισιόν. Πρώτα, για την περιφερειακή πολιτική, ίσως να μην κατενόησα καλά. Σημείωσα ένα νούμερο, ότι υπήρξαν εσφαλμένες πληρωμές της τάξης των 580 εκατομμύριων ευρώ. Και ε, μετά άκουσα και μια πρόταση, μια φράση δηλαδή σχετικά με την ανάκτηση των ποσών αυτών. Εκρεμεί αυτή η ανάκτηση. Πρώτα-πρώτα το αριθμητικό αυτό στοιχείο ήταν σωστό. Έχει γίνει ανάκτηση και σε ποιο βαθμό. Και μία ερώτηση ακόμα σχετικά. Πάει να πει αυτό ότι υπάρχει ακόμα μισό δισεκατομμύριο το οποίο επικρέμαται ως δαμόκλειο σπάθη επί των κεφαλών μας ε, ε, σχετικά με τον ελληνικό προϋπολογισμό. Δεύτερη ερώτηση για την Ευρωστάτ. Η δική μου εμπειρία μου λέει καλύπτει, καλύπτεται, ε, είναι ταυτόσιμη μάλλον με τις κυρίες Γκρέσλε. Ίσως είναι καθαρά γερμανικό πρόβλημα, αλλά όταν βγαίνει ο κόσμος και με ρωτάει η περίπτωση της Ελλάδας μας δείχνει ότι καλύτερα να είχαμε μείνει μόνοι μας, Φαίνεται πάντως μια σφαλμένη αντιμετώπιση των δειγμάτων που προμηνύουν κάποια κρίση. Και αυτό βέβαια θίγει την αξιοπιστία όλων των θεσμικών οργάνων. Εγώ υπεραμείνω με τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε τέτοιες περιπτώσεις λέγοντας, υπήρξε άλλωστε και ένα άρθρο στην γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung που έλεγε ότι και η Ευρωστάτ είχε επισημάνει την ανεπαρκή ποιότητα των ελληνικών ε, στατιστικών στοιχείων. Άρα πάει να πει ότι ο μηχανισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε καλά τη δουλειά του. Το Συμβούλιο Υπουργών γιατί δεν αντέδρασε. Μπορείτε να πείτε κάτι σχετικά με τι πολιτικέ αντιδράσει απέναντι ε, στι δικέ σας έγκαιρε προειδοποίησεις σχετικά με την ανεπάρκεια των στοιχείων. Τρίτο, έρχομαι σε αυτά που είπε ο Λιμπεράτης και πριν. διαβάζοντα τι εφημερίδε σημειώνω ότι η Ελλάδα δεν είναι η μοναδική χώρα που αντιμετωπίζει τέτοια τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα. Αναφέρονται και άλλες ε, χώρες μέλη, από ιδρυτικά μέλη μάλιστα της ε, ΕΟΚ, μέχρι και άλλες χώρες, οι οποίες πάντως είναι πολλά χρόνια μέλη. Διερωτώ που εν πάση περιπτώσει απέτυχαν οι μηχανισμοί ελέγχου Τη ε, Ένωση διότι αφενός υπάρχει το Σύμφωνο σταθερότητα, το οποίο προβλέπει μηχανισμούς ελέγχου. Μπορούμε να μιλήσουμε βέβαια για τι περιπτώσει προσπάθειας λύσεων και εκεί θα παίξει ένα ρόλο η Γερμανία, αλλά θα πρέπει να αποκλείονται από την αρχή οι κρίσεις και να μην φτάνουμε σε καταστάσει όχι όπω τη Ελλάδα μόνο, αλλά και άλλων χωρών. Τι έγινε λοιπόν, γιατί δεν εφαρμόστηκε ο μηχανισμός πρόληψης της κρίσης. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Οι κύριοι Γκάιερ και Λιμπεράτσκι έθεσαν ερωτήσεις. Μπορείτε να πείτε και κάτι σχετικά και σχετικά με τα μεγάλα ποσά που εμπλέκονται και για την πρόληψη επίση. Υπάρχουν κρίσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά οδυνηρές. Κάτι λοιπόν πρέπει να γίνεται και προληπτικά. Και εδώ βέβαια μέγα ρόλο μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Όλαφ πρώτα. Ο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι πρώτα ε, στα σχετικά με τη Γεωργία και το ΑΙΑΞ. Με ρώτησε η κυρία Γκρέσλε, έχετε κάποια επιφύλαξη. Ο κίνδυνος δεν ήταν χαρακτήρα δημοσιονομικού για την Ελλάδα. Αποκλείσαμε τη χρηματοδότηση ποσών που ήδη είχαν καταπέσει, εφόσον δεν επιλυνόταν οι προϋποθέσεις, για 620 εκατομμύρια ευρώ και άλλα 330 που βρίσκονται στην pipeline. Μιλούμε για 950 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είχαν αποκλειστεί από τη χρηματοδότηση. Ήταν περισσότερο κίνδυνος μείωση αξιοπιστίας τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια χώρα μέλου τη Ελλάδα, η οποία εξακολουθούσε μετά από μια δεκαετία να μην εφαρμόζει σωστά το σύστημα που ε, είχε συμφωνηθεί. Αυτό ήταν ο μεγάλο κίνδυνο. Όταν εν τέλει του 2009 εφαρμόστηκε ο μηχανισμός, είδαμε την επιφύλαξη. Τώρα, το περιθώριο σφάλματος λέει ότι είναι πάνω από 3%. Οι στατιστικές αποδεικνύουν το αντίθετο. Το περιθώριο σφάλματος είναι το random, που είναι 1,61. Συνολικά το περιθώριο σφάλματος μαζί και με τους ελέγχους στην βάση ανάλυσης κινδύνου, τότε φτάνουμε σε 3,9%. Δεν μπορεί όμως αυτό να, σε αυτό να γίνει η προβολή παρά μόνο στο random, δηλαδή 1,61%. Και ε, το νούμερο αυτό επιβεβαιώθηκε από το Certifying Body που επιβεβαιώνει τους λογαριασμούς και τις στατιστικές της Ελλάδας. Το τρίτο, για τον κύριο Λιπεράτσικη, τι μπορεί να γίνει δηλαδή για να ε, προ, όταν προμηνύονται τα, τα προβλήματα, αυτά που είπε ο Γενικό Μηδηθητή, σε αυτά θα δείτε μια κρίση σχετικά με τα συστήματα των διαφόρων χωρών, ανά χώρα, εάν δηλαδή είναι αξιόπιστοι οι μηχανισμοί του. Υπάρχουν, όταν υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, επιφυλάξει, θα δείτε ότι υπάρχει μια επιφύλαξη για το Ajax στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, που θεωρούμε ότι οι χώρε αυτέ δεν έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα ακόμα Επάρκω αποτελεσματικό. Και εξ ορισμού έχουμε φτιάξει ένα σχέδιο δράση μαζί με τις χώρες αυτές για να βελτιώσουμε την κατάσταση. σχετικά με την παρατήρηση ότι ίσως να οφείλεται το πρόβλημα στην ποιότητα των στατιστικών στοιχείων και έχουμε την, αν έχουμε την ικανότητα να προειδοποιούμε ε, για το ότι διαγράφεται η διακατάσταση, υπογραμμίζω και πάλι ότι η Ευρωστάτ περιορίζεται στη χορήγηση στατιστικών πληροφοριών. Η προτάσει της Κομισιόν σχετικά με την ενίσχυση των ε, οικονομικών ελέγχων Εμείς προτείνουμε στο Συμβούλιο να δώσει στην Ευρωστάτ την, ε, την ε, αρμοδιότητα αυτή έρευνας και για τις, στις επισκέψεις μεθοδολογικού χαρακτήρα όπου κάνουμε μια εξέταση εκτεταμένη όλων των στοιχείων. Περιοριζόμαστε ωστόσο στις στατιστικές πληροφορίες. Αυτός είναι ο στόχος της πρότασης. Να μπορούμε δηλαδή να περάσουμε και πέρα από τις στατιστικές πληροφορίες στην πηγή των πληροφοριών. Αυτός είναι ο στόχος της πρότασης που εκρήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, γιατί δεν λήφθηκαν υπόψη οι επιφυλάξεις της Ευρωστάτ. Η Ευρωστάτ πάντοτε τα τα πράγματα καθαρά. Από το 2005 η Ευρωστάτ έχει εκφράσει πέντε τουλάχιστον επιφυλάξει σχετικά με τα στατιστικά δεδομένα της Ελλάδας. Έχει κάνει δεκάδες αποστολών όλων των ειδών μεθοδολογικού χαρακτήρα διαλόγου ε, στην Ελλάδα. Άρα η ερώτηση αυτή μάλλον πρέπει να βεβαιωθεί στο Συμβούλιο και όχι στην Κομισιόν. Σημειώνω πάντως ότι είναι ε, θέματα τα οποία άπτονται ε, ενό διαρκού διαλόγου μεταξύ Ευρωστάτη και των, εθνικών, των ελληνικών εθνικών ε, στατιστικών αρχών. Αυτή είναι η απάντησή μου. Σε σχέση με την ε, περιφερειακή πολιτική, στο ερώτημα της κυρίας Γκρέσλε για τον προϋπολογισμό 2009 δεν υπήρχαν ε, επιφυλάξεις από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής. Απλώς δεν είχαν προχωρήσει τα προγράμματα. Επίσης διενεργήθηκαν έλεγχοι από τις ελληνικές αρχές καθώς και έλεγχοι από το ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο δεν βρήκε δυσλειτουργία του συστήματος ως προς τις συναλλαγές που έλαβαν χώρα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό καταρχήν. Επίσης θα ήθελα να πω ότι μετά από τις ε, διορθώσεις του 2005 οι Έλληνες ε, βελτίωσαν το σύστημα ελέγχου έτσι ώστε να μπορέσουμε να εχνηλατήσουμε στην πηγή τις ε, συστημικές ε, ασυνέπειες. Το 2009-2010, με βάση την απόφαση του 2005, οι ελληνικές αρχές προβαίνουν σε διόρθωση 10% σε όλες τις συμβάσεις δημόσιων έργων. Και αυτό μέχρι το τέλος του προγράμματος, το τέλος του τρέχοντος έτος. Αυτά όλα για να σας πω ότι υπάρχει ένας διορθωτικός μηχανισμός στην Ελλάδα που λειτουργεί, που και από πλευράς αρχών πιστοποίησης, και αρχών ελέγχου ως προς τα διαρθρωτικά προγράμματα και ταμεία. Άρα δεν μπορούμε να βάζουμε μαζί τις εισπράξεις που αφορούν την προγενέστερη περίοδο και τις πληρωμές οι οποίες εκταμιεύθηκαν για το 2010, δηλαδή ένα δις που καταβλήθηκε το 2009 για το οποίο δεν ανέκυψαν μεγάλα προβλήματα στο σύστημα. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις από πλευράς Επιτροπής, περνάμε στο τελευταίο τμήμα των διαδικασίων.